Mesdames et Messieurs, nous allons commencer. Nous sommes lundi, donc pas trop nombreux. και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα και δεν έχουμε πάρα πολλούς παρόντες όπως όλες τις Δευτέρες. Καλώς ήρθατε. Και θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης σημείωσε μια τροποποίηση στη μέση διάταξη. Ο κύριος Κάσμαν δεν μπορεί να μας παρουσιάσει το δικό του θέμα για την δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού στις 4 παρατέτατο όπως προβλέπετε, γιατί ακόμη δεν θα έχει φτάσει, είναι ακόμη στο αεροπλάνο. Ζήτησε λοιπόν να συζητηθεί το σημείο το δικό του τελευταίο στην ημερήσια διάταξη, γύρω στις 6 το απόγευμα, μετά τις παρουσιάσεις της Επιτρόπου Γεωργίευα και του Διευθυντού της ΦΑΟ, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω γιατί έδειξαν ευελιξία και δέχτηκαν αυτή την αλλαγή προγράμματος. Έχετε σχόλια, έχετε αντιρρήσει αν δεν έχετε αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη, όπως την τροποποιήσαμε. Έχετε λάβει και τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου του 2012. Αν έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά, παρακαλώ να τις δώσετε στη γραμματεία πριν το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά ως έχουν. Επίσης, στο φάκελό σας έχετε λάβει και τις συστάσεις και τις αποφάσεις από τις συνεδριάσεις συντονιστών της 22ης Ιανουαρίου. Αν έχετε παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίασης συντονιστών, παρακαλώ επίσης να τις αναφέρετε στη γραμματεία πριν το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. Διαφορετικά, τα αποτελέσματα αυτά θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν ως έχουν. Ωραία μουσική έχουμε βάλει. Άλλες ανακοινώσεις δεν έχω. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Ζητώ συγγνώμη αν μερικές φορές δεν είμαι απόλυτα συγκεντρωμένη σήμερα. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσεις. Δεν φαίνεται να έχει κάτι να μας ανακοινώσει η Επιτροπή. Έχουμε λάβει ένα ερώτημα από τον κύριο Ρικάρντο Κορτές Λάστρα προς την Επιτροπή. Το κείμενο το έχετε στο φάκελό σας. Ο κύριος Κορτές Λάστρα θέλει το λόγο? Όχι. Έχει κάποια απάντηση η Επιτροπή? Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ματία Σάλτμαν είναι το όνομά μου. Από τον τομέα ε, ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και θέλω να πω ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει το να προωθεί ε, το δίκαιο εμπόριο με διάφορα ε, εργαλεία και για το εμπόριο και για την εταιρική ευθύνη και για την αναπτυξιακή πολιτική για το εμπόριο, ίσως θα θυμάστε ότι έχουμε αναλάβει πολλές δεσμεύσεις ε, για να υποστηρίξουμε το δίκαιο εμπόριο και διάφορα προγράμματα ε, για τη βιωσιμότητα, για να βελτιώσουμε την ανάπτυξη Παραδείγματο χάρη υποστηρίζουμε διάφορα προγράμματα στις ε, κρατικές συμβάσεις και έχουμε μία ε, ανακοίνωση του 2011 για την εταιρική ευθύνη όπου επίσης αναφέρονται αυτά τα θέματα. Η ερώτησή σας περισσότερο στρέφεται για την, ε, γύρω από την πρόσφατη ανακοίνωσή μας όπου τονίζουμε τη σημασία της βιώσιμης γεωργίας και της αηφόρου γεωργίας στην ανακοίνωσή μας αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει η γεωργία σε μικρές εκμεταλλεύσεις και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σχετικό με αυτό το οποίο επιδιώκουμε και με το δίκαιο εμπόριο. Στο δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας ρωτάτε σε τι βαθμό, κατά πόσο υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ευαισθητοποίηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το δίκαιο εμπόριο. Στα εργαλεία που έχουμε για την αναπτυξιακή συνεργασία έχουμε ένα θεματικό πρόγραμμα για τις τοπικές αρχές για να εφαρμόζουμε προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για το δίκαιο εμπόριο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο για να προωθήσουμε το δίκαιο εμπόριο, όπως είπαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τα κράτη-μέλη προσπαθούμε να ε, τονίζουμε και να επενούμε τα κριτήρια δίκαιου εμπορίου στις κρατικές συμβάσεις. Παραδείγματο χάρη, ένα από τα σημεία, μία από τις προδιαγραφές για κάποιες κρατικές συμβάσεις μπορεί να είναι το δίκαιο εμπόριο. Και το τελευταίο τμήμα της ερώτησής σας με επαναφέρει στο θέμα της ε, ε, των θεμάτων που μας αφορούν για την ανάπτυξη και την αλλαγή. Και νομίζω ότι το δίκαιο εμπόριο είναι ένα από τα μοντέλα που έχουμε για την ανάπτυξη, γιατί είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ των παραγωγών του Νότου και των καταναλωτών του Βορρά και οι δύο πλευρές αντιπροσωπεύουν τον ιδιωτικό τομέα. Άρα εδώ έχουμε σαφώς ένα παράδειγμα όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να επιφέρει αλλαγή στον τομέα της ανάπτυξης. Άρα αυτά συμβαδίζουν με την προσπάθειά μας να δουλέψουμε στενά με τον ιδιωτικό τομέα και να ενισχύσουμε το ρόλο του ιδιωτικού τομέα για να επιτύχουμε τους στόχους της ανάπτυξης. Αυτά. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Cortés. Ευχαριστούμε. Κύριος Κορτές Λάστρα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή. Και ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή σε όλες τις πολιτικές, με συνέπεια, να έχει κατά νου το δίκαιο εμπόριο. Νομίζω ότι θα ακούσουμε και την παρουσίαση ε, του ΦΑΟ και θα δούμε ότι δεν είναι θέμα μόνο ποσότητας των τροφίμων που μπορούμε να παράγουμε, αλλά και θέμα διανομής των τροφίμων. Υπάρχουν τρόφιμα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες δίκαιου εμπορίου και μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ούτω ώστε αυτά τα τρόφιμα να διανέμονται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Θα ήθελα η Επιτροπή σε όλες τις πολιτικές της να συμπεριλαμβάνει το δίκαιο εμπόριο ακόμη και αναφέροντάς το. Είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε οικονομίες κλίμακος και για να υποστηρίξουμε τους μικρούς ε, παραγωγούς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει το λόγο. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Δεν κατάλαβα ότι ήταν ερώτηση, αλλά... Ναι, βεβαίως θα συμπεριλάβουμε όλα αυτά στις ε, εργασίες μας. Το κατάλαβα. Ωραία. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Άρα, για το επόμενο σημείο, κυρία Τζόρτζεβα, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, υποδεχόμαστε, ελπίζω να έρθει η κυρία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 Μπορείτε ευχαρίστω λοιπόν να κάνετε την ερώτησή σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το δίκαιο εμπόριο και για το πώς θέλετε να το επεξεργαστούμε στον ιδιωτικό τομέα. Πώς συμπεριλαμβάνει η Επιτροπή αυτό στις προτάσεις της για τις επιχειρήσεις τα 27 κράτη-μέλη. Πώς γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν οι εταιρείε ότι πρόκειται για κοινοτικό δίκαιο και αναφέρομαι σε μια εταιρεία παραδείγματο χάρη η οποία βρίσκεται στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία και συνεργάζεται παραδείγματο χάρη με την Τζακάρτα. Πώς ενημερώνεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, για ό,τι έχει σχέση με την δεοντολογία και για τα εθελοντικά αυτά προγράμματα δεν έχουμε, αν θέλετε, δυνατότητα να τα επιβάλλουμε. Πρόκειται για ένα σύστημα προαιρετικό. Το μόνο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε αυτούς που εργάζονται στο σύστημα αυτό έτσι ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και αυτό βεβαίως μέσω των διαφόρων προγραμμάτων. Αυτό πολύ συγκεκριμένα για τα προγράμματα στην Ινδία. Στηρίζουμε, χρηματοδοτούμε τα προγράμματα αυτά και άλλα που αφορούν το δίκαιο εμπόριο, έτσι ώστε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτές. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, τίποτα παραπάνω, γιατί επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει, αν θέλετε, ένα πρότυπο που πρέπει να επιβληθεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε σε επιχειρήσεις πρέπει να επιβάλλετε ή να υιοθετήσετε αυτά τα πρότυπα για το δίκαιο εμπόριο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, πολλές επιχειρήσεις και πολλά πρότυπα. Πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς. Υπάρχουν πολλαπλά συστήματα υποστήριξης του δίκαιου εμπορίου και ε, το σημαντικό είναι να βρεθούν οι εταίροι στον ιδιωτικό τομέα που θα συνεργαστούν στη βάση αυτών των αρχών. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο, στο επόμενο σημείο με μεγάλη χαρά. Καλωσορίζουμε την Επίτροπο Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Είναι πολύ σοβαρές, όπως ξέρετε, οι συνθήκες που μας απασχολούν σήμερα στο Μάλι και στην ε, Συρία. Πολύ σοβαρές και λίγες είναι οι ελπίδες μας όσον αφορά τη Συρία. Κυρία Επίτροπε, μας επισκεφτήκατε το Δεκέμβριο και ήδη είχατε αναφερθεί στην κρίση στο Μάλι και στη Συρία. Για το Μάλι είχατε πει ότι ανησυχείτε ότι η κρίση η πολιτική είναι πολύ σοβαρή. Ο εξτρεμισμός χαρακτηρίζει πολλές από τις συνιστώσεις της κοινωνίας στο Μάλι. Σήμερα είδαμε την στρατιωτική επέμβαση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων και τις αφρικανικές δυνάμεις μίσμα που στηρίζουν αυτήν την επιχείρηση καθώς και την στήριξη στις ε, ένοπλες δυνάμεις στο Μάλι από μέρους άλλων ε, χωρών. Ξέρουμε επίσης ποιες είναι οι συνέπειες, οι άμεσες για τους πιο ευάλωτους ε, πολίτες. Ξέρω ότι επισκεφτήκατε την περιοχή πολύ πρόσφατα και με μεγάλη ανυπομονησία θα σας ακούσουμε. Μετά από δύο χρόνια βίας, η κατάσταση στη Συρία παραμένει πάρα πολύ ανησυχητική. Σήμερα δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τους πολίτες της Συρίας και άλλους. Βεβαίως σήμερα γνωρίζουμε ότι ο διάλογος με το καθεστώς του Μπασάρ Ελασάντ έχει διακοπεί η έκρηξη που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στα σύνορα της Συρίας και της Τουρκίας μας έδειξε πόσο σοβαρή παραμένει η κατάσταση. Θα σας ακούσουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά και ξέρουμε ότι σήμερα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αυτοί που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και οι άλλοι, βρίσκονται επί τόπου και θεωρούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας ενημερώσω σχετικά με τις εξελίξεις ε, στο Μαλί και στην Συρία, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ε, είδαμε σημαντικές εξελίξεις ε, στη μία περίπτωση προς το καλύτερο και στην άλλη προς το χειρότερο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την περίπτωση όπου είδαμε εξελίξει προς το καλύτερο, ε, αν και μας περιμένουν σημαντικές δυσκολίες. Ε, η περίπτωση αυτή είναι το Μαλί. Στην ε, Επιτροπή σας, μετά από ταξίδι στο Μάλι, φοβούμουν πολύ ότι η κατάσταση στο Βορρά ε, ήταν πολύ δύσκολη και ότι από ε, ανθρωπιστικής πλευράς ε, δημιουργούνταν εντάσεις ε, και στις γειτονικέ χώρες. Γι' αυτό ένιωσα ανακούφιση που η Γαλλία αποφάσισε να παρέμβει και στις 22 Ιανουαρίου. Επισκέφτηκα και πάλι το Μπαμακό για να έχω από πρώτο χέρι εικόνα σχετικά με το τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και κατόπιν με τον Υπουργό επισκεφτήκαμε ε, πρόσφυγες από το Μαλί. Ε, σήμερα μάλιστα ε, συναντήθηκα για δεύτερη φορά με τον ε, αναπληρωτή πρωθυπουργό του Μάλι και Μιλήσαμε για τη δυνατότητα της χώρας να αλλάξει ε, τη μοίρα της χώρας, να ε, επιστρέψει στη δημοκρατία με εκλογές και με στρατιωτική παρέμβαση να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στο Βορρά. Σύντομα, να σας ε, αναφέρω τι συμβαίνει στο ανθρωπιστικό μέτωπο και τι μας περιμένει. Καταρχήν, η ανθρωπιστική κατάσταση στο Μάλι, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, ε, συνεχίζει να είναι δραματική. Βλέπουμε για μια χώρα που έχει χτυπηθεί από αλλεπάλληλες κρίσεις. Είχαμε κρίση τροφίμων πέρσι, είχαμε την πολιτική και τώρα ε, τη σύγκρουση στο βορρά ευάλωτοι πληθυσμοί. Ε, βλέπουμε ότι είναι ε, δεύτερη σε παιδική θνησιμότητα σε παιδιά ε, κάτω των 5 ετών μετά τη Σομαλία. Η σύγκρουση έχει δημιουργήσει μεγάλο αριθμό προσφύγων στις γειτονικές χώρες. 167.000 την προηγούμενη εβδομάδα και 227.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι στο νότο, στον Πάμακο και γενικά στο νότο του Μάλι μετά την 11η ε, Ιανουαρίου έχουν ε, αυξηθεί εσωτερικά ε, εκτοπισμένοι, αλλά κατά σχετικά μικρούς αριθμούς 22.000 περισσότεροι κατοχωρημένοι πρόσφυγες σε σχέση με πριν την 11η Ιανουαρίου και 4.000 ε, παραπάνω εσωτερικά ε, εκτοπισμένοι. Δεν ε, είμαι βέβαιη για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, αλλά υπάρχει εκτοπισμός ανθρώπων, αλλά όχι σε τόσο σημαντικό βαθμό. Αυτό που μας απασχολεί είναι ότι δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε όσον αφορά ε, τους ε, εκτοπιστέντες και τους πρόσφυγες. Ε, δεν ξέρουμε αν μπορεί να έχουμε κάποιο γεγονός το οποίο να οδηγήσει περισσότερους ε, στην προσφυγιά, για παράδειγμα εθνοτικές εντάσεις ή μήπως ε, μας περιμένει το αντίθετο, μαζική επιστροφή, κάτι που θα δημιουργήσει ε, εντάσεις όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση στον βορρά του Μάλι. Τρία πράγματα γνωρίζουμε. Καταρχήν, δεν Το πρόβλημα δεν είναι η αύξηση των αναγκών, είναι η πρόσβαση στο βορρά. Μετά την επίσκεψή μου στις 22 Ιανουαρίου, ζητήσαμε να δοθεί περισσότερη προσοχή στην παροχή δυνατότητας ε, των ε, ε, ανθρώπων των ανθρωπιστικών οργανώσεων να μετακινούνται στο βορρά της χώρας. Αλλά Είναι ζωτική σημασία να ανοίξουμε περισσότερες δυνατότητες ε, για την ε, παράδοση προϊόντων στο βορρά. Επίσης, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν νέε απειλέ, Για παράδειγμα, νάρκες και εκρηκτικές ύλες έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στις παραδόσεις αγαθών. Και τρίτον, Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ανάγκες και στο νότο της χώρας και σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε τον νότο της χώρας ε, και τις ε, άμεσα γειτονικές περιοχές. Έχουν αυξηθεί και εκεί οι ανάγκες. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακεφαλαιώσω. Η Κομισιόν ε, είναι ο σημαντικότερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας μέχρι τώρα. Έχουμε δώσει 93 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό το ανακοίνωσα κατά την ε, τελευταία μου επίσκεψη εκεί. Ε, στα 93 εκατομμύρια ε, συμπεριλαμβάνονται και 15 εκατομμύρια επίγουσας βοήθειας ε, μέσω του Ταμείου ε, Ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα χρήματα προέρχονται από την ΕΚΟ. Θα ανακοινώσουμε επιπλέον 22 εκατομμύρια. Έτσι το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 115 εκατομμύρια ευρώ και είναι πολύ πιθανό να πρέπει να διαθέσουμε περισσότερους πόρους τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας. Ε, για την επίγουσα ανάγκη, διότι θα χρειαστεί να χτυπήσουμε την πόρτα σας ε, για να χρησιμοποιήσουμε ε, το αποθεματικό για την επίγουσα βοήθεια. Τι κάνουμε. Προσπαθούμε να καλύψουμε βασικές ανάγκες των προσφύγων στον Ήγηρα, στην Πουρκίνα Φάσο και τη Μαυριτανία. Νερό, στέγαση και καταλήματα και ε, εγκαταστάσεις υγιεινής, ε, βοηθάμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, να διατηρήσουν ε, τις ε, βασικές υπηρεσίες στους ανθρώπους στον βορρά του Μάλι παρά τις πολύ σκληρές συνθήκες. Το 18% των καταβλισμών στο βορρά συνεχίζει να λειτουργεί χάρη στη βοήθειά μας μετά την περσινή κρίση. Μετά την κρίση βοηθήσαμε και στη διατήρηση της παροχής νερού στον Τιμπουκτού. Επιτρέψαμε στον Ερυθρό Σταυρό να, δώσει, να παράσει τροφική βοήθεια 150.000 ε, ανθρώπου στο βορρά του ε, Μαλή. Έχουμε βοηθήσει στην παροχή υπηρεσιών στους ε, εσωτερικά εκτοπισμένου στο νότο του Μάλι. Και τέλος, είμαστε παράγοντα κλειδί για την καταπολέμηση της, του υποσυτισμού. 50.000 παιδιά πάσχουν από οξύ υποσυτισμό εμείς λοιπόν ε, βοηθάμε ε, στις περιπτώσεις αυτές ε, και βέβαια δεν είναι μόνο τα χρήματα σημαντικά. Συνεργαζόμαστε συνεχώς με τον ΟΗΕ, με τον Ερυθρό Σταυρό για να αξιολογήσουμε τις ανάγκες, να ζητήσουμε, να επιστήσουμε την προσοχή του κόσμου στις ανθρωπιστικές δράσεις. Τι Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα θα είναι να έχουμε μια, ένα ομαλό πέρασμα από την επίγουσα βοήθεια σε γρήγορη επανεκκίνηση της αναπτυξιακής βοήθειας ε, και την ε, αποκατάσταση της διακυβέρνησης ε, στο σύνολο της χώρας και ιδιαίτερα στο Βορρά. Αυτό το συζητήσαμε με τους Υπουργούς Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο την προηγούμενη εβδομάδα ο συνάδελφος μου Πίμπαλξ ανακοίνωσε ότι ε, επανερχόμαστε στην ε, αντιστοιχική βοήθεια ε, στο Μαλί 215 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν και με προϋπόθεση η χώρα να προοδεύσει στην ανοικοδόμηση των θεσμών της χώρας. Επίσης, ε, πολύ σημαντικό είναι να, ξεκινήσουν, να ξεκινήσει πάλι η παροχή δημοσίων υπηρεσιών ε, στο Τιμπουκτού, για παράδειγμα, και αλλού. Ε, οι υπηρεσίες αυτές διακόπησαν πολύ απότομα κατά τη διάρκεια τη κυβέρνηση εξουσίας των Ισλαμιστών στο Βορρά. Ιδιαίτερα θέλουμε να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές ε, να ε, ανοικοδομήσουν τις ε, διάφορες δομές στο βορρά. Με τον Επίτροπο Πίμπαλξ αυτό που προσπαθούμε είναι να γεφυρώσουμε να δημιουργήσουμε σύνδεσμο ανάμεσα στις, ε, στην ε, επίγουσα βοήθεια και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Βοηθούμε δηλαδή τις ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, να επιταχύνουν ε, την ανοικοδόμηση των δομών και έχουμε μια πολύ καλή εταιρική σχέση για το μεταβατικό αυτό στάδιο στην ακτή Ελεφαντοστούν λαμβάνοντας εκμεταλλευόμενη την τοπική παρουσία ε, των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ώστε να παράσουμε βοήθεια διάσωσης, αλλά να ε, έχουμε και μετάβαση προς την ανάπτυξη. Και έτσι θα μπορέσουμε πιο γρήγορα να δούμε ανάπτυξη. Πέρα από την ανθρωπιστική κατάσταση, ε, θα έχετε ακούσει πολύ ανησυχητικές ε, αναφορές σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ιδιαίτερα έχουμε δει φόνους από εκδίκηση και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, έχουμε συζητήσει με τις ε, αρχές στο Μάλι, ε, το έχω συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτρέψουν οι εθνοτικές εντάσεις να πλήξουν το βορρά του Μάλι. Εγώ δεν γνώριζα καλά τη χώρα. Κατά τις, επισκέψεις, τις πρόσφατες επισκέψεις μου έμαθα πολλά πράγματα. Ε, ναι, έμαθα ότι οι άνθρωποι στο βορρά και στο νότο ε, δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα. Ε, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα, εκτός αν επικεντρωθούμε στο πρόβλημα αυτό. Είπα σήμερα στον Πρωθυπουργό ότι έγιναν φρικτά πράγματα στο Βορρά, αλλά αυτός, αυτό δεν θα πρέπει ε, να είναι αιτία να γίνουν ε, ακόμα περισσότερα φοβερά πράγματα. Ε, στην Ευρώπη μπορούμε να είμαστε περήφανοι που θεωρούμε τον σεβασμό του ε, διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ως κεντρικό θέμα και θα πρέπει ο στρατός μεν να μπορεί να πολεμήσει αλλά να μπορεί να προστατεύσει ε, και τους ε, πολίτες και να βοηθήσει στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ελπίζουμε ότι θα γίνει προσεκτική αξιολόγηση της κατάστασης από τη Γαλλία όσον αφορά τη δική της παρουσία εκεί, διότι ναι, είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας εκεί όμως. Δεν θα πρέπει να γίνει η πρώιμη απόσυρση των στρατευμάτων. Επίσης, γνωρίζουμε ότι εντάσεις αιώνων δεν μπορούν να ξεχαστούν γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επενδύσουμε σε μέτρα συμφιλίωσης ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. Αυτό όμως ε, θα είναι κάτι πολύ μακροπρόθεσμο. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις άλλες χώρες ε, της ζώνης Σαχέλ. Συνεχίζουμε και εκεί τις προσπάθειές μας και όπως ξέρετε θέλουμε να βοηθήσουμε στην ε, αντίσταση κατά των φυσικών καταστροφών ε, στην ε, ζώνη Σαχέλ. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, την υποστήριξή μας προς τη ζώνη Σαχέλ και μακροπρόθεσμα. Και βέβαια βασιζόμαστε σε εσάς εδώ στο Κοινοβούλιο ε, να ε, συνεχίσετε να μας βοηθήσετε στην υποστήριξή μας στη ζώνη Σαχέλ. Να προχωρήσω τώρα στη Συρία όπου δυστυχώς ε, τα πράγματα έχουν πάει από το κακό στο χειρότερο μετά την τελευταία μας συνάντηση στις 18 Δεκεμβρίου. 430.000 πρόσφυγες είχαμε όταν ήρθα εδώ 600.000 πέρασαν τα σύνορα ε, τον Ιανουάριο, τώρα ε, ανέρχονται σε 830.000. Και αυτό σημαίνει ότι ε, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα ξεπεράσουμε το όριο του 1 εκατομμυρίου προσφύγων. Ε, η κατάσταση είναι κακή λοιπόν ε, και για τους πρόσφυγες ε, και για τις γειτονικές χώρες. Είναι ακόμα χειρότερη όμως η κατάσταση μέσα στη χώρα όπου οι διαμάχες δυσκολεύουν την παροχή βοήθειας προς τους ευάλωτους και αποδυναμωμένους ανθρώπους. Στον χάρτη, εδώ από πίσω μου βλέπετε πού μπορούμε να παράσχουμε βοήθεια πού μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια σε τακτική βάση, πού είχαμε κάποιες ε, επιτυχίες, ε, αλλά και πού συναντάμε σημαντικές δυσκολίες και πού ουσιαστικά δεν έχουμε καμία πρόσβαση. Υπάρχουν ε, περιοχές όπου ε, έχουμε ε, πρόσβαση χωρίς προβλήματα. Είναι οι πράσινε περιοχέ, αλλά δυστυχώ αυτή η περιοχή συρρυκνώνεται και είναι ήδη μικρή. Ε, κίτρινες είναι οι περιοχές όπου ε, έχουμε μερικές φορές πρόσβαση, όχι όμως σε τακτική βάση και κόκκινες είναι οι περιοχές όπου η κατάσταση είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Προφανώς λοιπόν ε, ε, μεγάλο μέρος της βοήθειας δεν φτάνει τους ανθρώπους ε, εντός της Συρίας και αυτό οδηγεί και τους ανθρώπους να φύγουν, να περάσουν τα σύνορα. Θέλω όμως επίσης να σας πω και αυτό δείχνει ο χάρτης ότι όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση δεν ήταν αδύνατο να παράσουμε βοήθεια Λέγεται κατά καιρού ότι η βοήθεια παρέχεται μόνο σε περιοχές ε, που ελέγχονται από την κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν αληθεύει. Να σας δώσω τρία παραδείγματα του πώ χρηματοδοτούμε την παροχή βοήθειας στο βορρά της Συρίας, σε περιοχές που ελέγχονται ε, ε, από τους από τους ε, ε, έχουμε παράσχει ε, πακέτα υγιεινής στην περιοχή Homes. Ο UNHCR έχει φτάσει και στην περιοχή Αζάς, στο Αλέπο, στον βορρά της Συρίας, παρέχοντας σκηνές κλπ. Είχαμε μια ε, εκστρατεία με αεροπλάνα, πέντε αεροπλάνα ε, στην Λατάκια και ε, ένα κονβόι 8 φορτηγών προς το Αζάζ. Δεν ξέρω αν βλέπετε τις περιοχές αυτές στο χάρτη. Είναι περιοχές λοιπόν που ελέγχονται και από, τους, και από την κυβέρνηση και από τους εξεγερθέντες. Δεύτερο παράδειγμα, ε, στις 15 ε, Φεβρουαρίου η ε, αποστολή του ΟΗΕ παρέδωσε κάποια αγαθά σε 6.000 εσωτερικά εκτοπισμένους στο Καραβέ βορειοδυτικά, στα βορειοδυτικά της Συρίας στην περιοχή Ιτλίπ. Και Επίσης, αποστέλλεται περισσότερη περιοχή σε 25.000 ε, ανθρώπους. Επίσης, ε, χρηματοδοτούμε μια μη κυβερνητική οργάνωση που βοηθάει 15.000 ανθρώπους που έχουν κολλήσει στα, στους καταβλισμούς. Στο ΑΡΠΕΙ έχετε ακούσει για τους καταβλισμούς αυτούς ε, στο σύνολο με την Τουρκία, αλλά εντός της Συρίας. Και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε περισσότερα εφόσον οι γειτονικέ χώρες επιτρέψουν στους εταίρους μας να κάνουν περισσότερα. Αυτή διαδικασία όμως δεν είναι εύκολη και απλή. Συνεργαζόμαστε στενά με το Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με ε, τον Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων της Τουρκίας και Οικογενειακών Υποθέσεων και συζητήσαμε πώς μπορούμε να ε, αυξήσουμε την ευρωπαϊκή βοήθεια, τι μπορεί να κάνει η Τουρκία ώστε να μας βοηθήσει να κάνουμε περισσότερα για τους Σύριους που βρίσκονται στην Τουρκία. Εγώ πρότεινα να έχουμε ένα νέο καταβλισμό χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όμως να συμμετέχουμε ε, από την αρχή στο σχεδιασμό και θα πρέπει να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε τα δικά μας κανάλια, ε, δηλαδή ε, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, που είναι οι εταίροι μας. Είχαμε μια πικρή επιτυχία, θα έλεγα, στο Κουβέιτ, ε, σε μια διάσκεψη ε, χορηγών, διότι η επιτυχία, επειδή 1,5 εκατομμύρια δολάρια ζήτησε η διάσκεψη αυτή για το επόμενο εξάμεινο, πικρή ήταν η επιτυχία όμως, και επιτυχία επειδή ε, λάβαμε το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ήταν πικρή η επιτυχία αυτή, διότι... Πρόκειται για μια κρίση που μπορεί να λυθεί μόνο με πολιτικά μέσα και ε, δεν βλέπουμε ακόμα ε, την επίτευξη του στόχου μας. 272 εκατομμύρια ευρώ έχει υποσχεθεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το μεγαλύτερο ποσό, ε, και είμαι πολύ περήφανη που η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη μαζί υποσχέθηκαν να δώσουν το ποσό αυτό. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Σουηδία και Γέρμανη είναι οι χώρες ε, που ε, διέθεσαν τα μεγαλύτερα ποσά, αλλά και πολλές άλλες χώρες ε, έχουν υποσχεθεί χρήματα. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι και πάλι ευρωπαϊκή υποστήριξη. Και το ποσό αυτό προστίθεται στα 323 εκατομμύρια που ήδη έχουμε διαθέσει αλλά ακόμα και αυτά τα σχεδόν 600, ευρώ, 600 ε, εκατομμύρια ευρώ δεν ε, θα ε, είναι το σύνολο της ανθρωπιστικής μας βοήθειας. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει και πάλι να αυξήσουμε τη βοήθειά μας προς τη Συρία. Όσον αφορά τη Συρία θα ήθελα να κλείσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε να πολιτικοποιούμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Ε, οι πυροβολισμοί κατά των ε, νοσοκομιακών ε, και των κονβόι βοήθειας είναι πάρα πολύ ε, ε, προβληματική, διότι ε, θα πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην λέμε ότι θα βοηθήσουμε τους εξεγερθέντες και γι' αυτό θα σας δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια ή να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Η ουδετερότητα και η αντικειμενικότητα θα οδηγήσει στη διάσωση περισσότερων ζωών. Αυτά δεν είναι απλά λόγια, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι κάτι που το βλέπω κάθε μέρα, διότι η πολιτική λύση δεν θα βρεθεί ε, πληρώνοντας τους πολιτικούς και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Είναι λοιπόν μεγάλος ο πειρασμός ε, να πολιτικοποιήσουμε το θέμα αυτό. Θα πρέπει όμως ε, να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι κάτι τέτοιο δεν θα βοηθήσει κανέναν. Δεν θα βοηθήσει την εξέβρεση πολιτικής λύσης. Θα χάσουμε ουσιαστικά ε, το μόνο μας εργαλείο που είναι που αποτελεί μια πραγματική ανάγκη να βοηθήσουμε ανθρώπου. Θα ήθελα και όσον αφορά το Μάλι και όσον αφορά τη Συρία, θα ήθελα να γνωρίσω την συμβολή του προσωπικού μας, του προσωπικού της ΕΚΟ, που έχει δώστε τη δυνατότητα στην Ευρώπη να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Και τώρα τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να πάρουν το λόγο. Θα ξεκινήσω εγώ. Μια ερώτηση που αφορά τους ε, μετατοπιστέντες και κυρίως τα νεαρά κορίτσια, τα οποία πολλές φορές αναγκάζονται να ε, προσθέξουν στην ε, πορνεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τι γνωρίζετε γι' αυτό. Ο κύριος Μπέρκμαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο για αυτήν την ε, παρουσίαση που μας έκανε για το Μάλι και για τη Συρία. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσει την ε, ευγνωμοσύνη του και το θαυμασμό για το ανθρωπιστικό έργο το οποίο έχετε αναλάβει και αυτά που προσφέρετε στους πολίτες της περιοχής του Μάλι και της Συρίας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει κανείς τα προβλήματα και την ανασφάλεια στο βόρειο τμήμα του Μάλι. Ήμουν στη Washington την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί μίλησα με πολλούς ε, με τον Τζόνι Κάρσον και με τον φαντάζομαι το γνωρίζετε υπεύθυνο στο Υπουργείο Εξωτερικών ε, των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα Αφρικής αλλά και με πολλούς από την Παγκόσμια Τράπεζα και πιστεύω ότι πραγματικά αυτό που σήμερα επήγει είναι η διακυβέρνηση να ενισχυθεί στο Μαμάκο και να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ενότητα της χώρας. Η ανθρωπιστική βοήθεια βεβαίως και κατόπιν αυτό που είναι το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη, η αναπτυξιακή βοήθεια έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να αποφευχθεί η διάσπαση του κράτους και οι αποσχιστικές ε, τάσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Ποια είναι η ανάλυση σας όσον αφορά τις πιθανότητες για μια ενίσχυση της ε, διακυβέρνησης από μέρους της πρωτεύουσας. Ξέρω ότι έχετε κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες, ότι συναντήσατε επί τόπου την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τι έχετε να πείτε για τις εκλογές μέσα στο 2013 που είναι ίσως η προϋπόθεση για να υπάρξει στήριξη, στήριξη παραδείγματος χάρη από τις Ηνωμένε Πολιτείες οι οποίοι δεν μπορούν να στηρίξουν αν ε, υπάρξει πραξικόπημα. Και έχετε να πείτε λοιπόν, ξέρω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιους ενδιασμούς όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση στο Μάλι. Επίσης, όσον αφορά την στρατιωτική επιχείρηση, ξέρουμε τι συμβαίνει ε, με την Αλκάιδα και ξέρουμε ότι συνεχίζουν να υπονομεύουν την κατάσταση στο Μάλι και κυρίως στο βόρειο τμήμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαρτίνες Μαρτίνες για την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση, αλλά ήθελα να πάρω το λόγο για να πω ότι σήμερα Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον ε, γεύμα με τον Πρωθυπουργό του Μάλι και κάποια μέλη του Κοινοβουλίου ήταν παρόντες μέλη της Επιτροπής μας και πραγματικά ακούσαμε τις απόψεις τους και εδώ θα ήθελα πραγματικά να πω ότι οι ευχαριστίες μας για όλα τα όσα έχετε κάνει είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές και θα πρέπει να τις επαναλάβουμε. Εγώ ήμουν στην ε, συνέλευση των ε, χωρών της Αφρικής, Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλήσαμε για το θέμα της IT. Ε, Έχουμε εξετάσει την κατάσταση εκεί και με μεγάλη ικανοποίηση θα ήθελα να σας πω ότι ακούγοντας τα πολύ ενθαρρυντικά λόγια για την κατάσταση στη χώρα αυτή, θα πρέπει πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε κύριε Επίτροπε για τα όσα κάνετε και αυτό αντιστοιχεί σε όλα όσα μας έχουν ε, πει και οι πρέσβεις μας εκεί επιτόπου στον Άγιο Δομήνικο, και στο υπόλοιπο τμήμα του νησιού. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όλα όσα κάνετε κυρία Επίτροπε και για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας πω ότι για μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο να ακούμε ότι το έργο σας αναγνωρίζεται, το δύσκολο έργο σας αναγνωρίζεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Όλοι μιλούν με μεγάλο σεβασμό για το έργο σας στην IT αλλά και αλλού στον κόσμο. Και γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ θετικό και ήθελα να το αναφέρω εδώ ενώπιον σας. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Θα αρχίσω με την απάντηση στην ερώτησή σας. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα όταν υπάρχουν εσωτερικές εκτοπίσεις, όταν υπάρχουν στρατόπεδα, και καταβλισμοί. Η προστασία πάντοτε αποτελεί πρόβλημα. Και ποιοι υποφέρουν περισσότερο, οι γυναίκες. Και το βλέπουμε σε όλους τους ε, καταβλισμούς. Και η κατάσταση των προσφύγων στη Συρία. Ακούμε σχετικές ιστορίες ότι παντρεύονται τα κορίτσια με πλουσίους, που στην ουσία σημαίνει ότι πουλιούνται σε πλουσίους. Ε, είναι εξαναγκασμένη πορνεία αυτό το οποίο γίνεται. Προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε μέτρα προστασίας, μέτρα που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των ευάλωτων ατόμων ε, και εδώ συμπεριλαμβάνονται και το πώς χτίζονται οι καταβλισμοί προσφύγων και το τι προστασία παρέχουμε στις γυναίκες και τι δυνατότητες τους δίνουμε να εκφραστούν. Αλλά το πρόβλημα παραμένει και είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε με ειλικρίνεια. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τις γυναίκες σε αυτούς τους καταβλισμούς είναι να δώσουμε κάποια ελάχιστη ευκαιρία απασχόλησης σε αυτές τις γυναίκες, γιατί αυτό θα τους δώσει αξιοπρέπεια, ε, τις κάνει περισσότερο ορατές και πολύτιμες. Στην Μπουρκίνα Φάσο με τον Γάλλο Υπουργό που ήμουν εκεί, έμαθα κάτι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες του ΑΡΕΓ. Ότι οι γυναίκες του ΑΡΕΓ είναι αυτές που φέρουν ε, το βάρος ε, της ευθύνης της εργασίας στην οικογένεια και αυτό το είχα ακούσει. Το χειρότερο όμως για αυτές που βρίσκονται σε στρατόπεδα προσφύγων ε, είναι ότι δεν μπορούν να δουλέψουν και αποτελούν κακό παράδειγμα για τα μικρά κορίτσια. Μου είπαν λοιπόν οι γυναίκες βοηθήστε μας, όχι μόνο για να βοηθήσετε μας προσωπικά, βοηθήστε μας για να μάθουμε στα κορίτσια μας, στις κόρες μας να δουλεύουν. Διαφορετικά ε, ε, στην κοινωνία θα είναι χαμένες ε, στην χώρα μας. Και τους έδωσα μια υπόσχεση. Να, βλέπω και τον συνάδελφο τον Κιμ που ήμασταν μαζί στην αποστολή αυτή. Υποσχεθήκαμε ότι θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να δουλέψουν σε διάφορες εργασίες χειροτεχνίας τους καταβλισμούς και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο γιατί δεν είναι κάτι που τους σώζει τη ζωή, αλλά από την άλλη πλευρά είναι αλήθεια ότι όντως τους σώζει τη ζωή το να έχουν κάποια απασχόληση και είναι πολύ σημαντικό να το προωθήσουμε. Και να πω και κάτι ακόμη για τους πρόσφυγες ε, του Μάλι είναι νομαδικοί λαοί, είναι άνθρωποι που μετακινούνται πολύ εύκολα και μπορούν εύκολα να μαζέψουν ε, τα υπάρχοντά τους και να μετακινηθούν. Μετακινούνται λοιπόν από την άλλη μεριά των συνόρων. Πάνε στην Μπουρκίνα Φάσο, φτωχή χώρα. Στον Ήγηρα, φτωχή χώρα. Στη Βαβριτανία, επίσης φτωχή χώρα και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ηθικά σωστό γιατί τους βοηθάμε. Τους βοηθάμε με τρόφιμα, με εκπαίδευση, με φαρμακευτική περίθαλψη, αλλά βοηθώντας τους, τους δημιουργούμε έναν παράγοντα που τους έλκει να μείνουν εκεί. Άρα επεμβαίνουμε στις συνήθειές τους. Και συζητούσαμε τον Κιμ σήμερα ότι έχει κέρια σημασία να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον επαναπατρισμό. Δηλαδή, να φροντίσουμε οι συνθήκες μέσα στο Μάλι να είναι εξίσου καλές με τις συνθήκες στον καταβλισμό προσφύγων. Όταν βρίσκονται λοιπόν οι πρόσφυγες σε καταβλισμού, να φροντίσουμε να υπάρχουν συνθήκες αξιοπρέπειας και περίθαλψης και ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτου και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργούμε και συνθήκες επιστροφής στον τόπο τους για να μην μένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στου καταβλισμού προσφύγων. Προ τον κύριο Μπέρμαν τώρα. Είμαι σχετικά αισιόδοξη ότι θα γίνουν εκλογέ στο Μάλι Νομίζω 31 Ιουλίου ήταν η ημερομηνία που είχε δοθεί. Και οι εκλογές αυτές ελπίζουμε να είναι σχετικά επιτυχημένες και να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη στη χώρα. Θα συνεχιστεί όμως η σκληρή δουλειά που απαιτείται μετά τις εκλογές, γιατί θα πρέπει μετά τις εκλογές να υπάρξουν και θεσμοί παντού και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί το ξέρουμε ότι το Μάλι ε, πλήγει πάρα πολύ από το πραξικόπημα, διότι το πραξικόπημα δεν σήμανε μόνο ότι έφυγε από τη θέση του ο πρόεδρος και υπήρχαν κάποιοι αξιωματικοί που είχαν παράνομα την εξουσία. Το πραξικόπημα σήμανε και λαιλασίε. Εκλάπησαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καταστράφηκαν αρχεία σε κυβερνητικούς φορείς. Και το πραξικόπημα επίση σημαίνει ότι αυτοί που βρίσκονταν σε θέσει εξουσίας δεν βρίσκονται πια σε αυτές τις θέσεις και δεν υπάρχει κάποιος άλλος πόλος βαρύτητας. Ε, και όταν ρωτάω ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Μάλι, ποιος είναι ο διαφαινόμενος ηγέτης, δεν είναι καθόλου σαφές. Επομένως, αποκατάσταση της αρχής θα υπάρξει, αλλά θα είναι μια μακρά διαδικασία αυτή και θα πρέπει να επενδύσουμε στη δημιουργία θεσμών και για μεγάλο διάστημα μετά τις εκλογές. Επίσης πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το ότι οι εκλογές θα φέρουν στην εξουσία κάποιους που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη για να ενώσουν τη χώρα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος, αλλά ο οποιοδήποτε πρόεδρος μάλλον θα χρειαστεί περισσότερη υποστήριξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για την IT. Πήγα για την τρίτη επέτειο ε, Και όταν έφυγα, να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι θα ήταν φρικτή η κατάσταση, γιατί η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα αρνητική και εξεπλάγει, διότι η κατάσταση είναι καλύτερη Ίσως γιατί περίμενα τα χειρότερα. Τέλος πάντων είναι καλύτερη κατάσταση από ό,τι ανέμενα. Ε, καταρχήν διότι έχει γίνει πολλή δουλειά για την αποκατάσταση μετά το σεισμό, πολύ περισσότερη δουλειά από ό,τι ακούμε. Από τα 1,6 εκατομμύρια που έχασαν τα σπίτια τους, το 1,2 εκατομμύρια βρίσκονται σε, έχουν κάποια στέγαση. Και δεύτερον, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά με αυτή την προσπάθεια έδειξε τι μπορούμε να κάνουμε με εντυπωσιακό τρόπο. Το Κοινοβούλιο μας επέστησε την προσοχή, μας είπε να το προσέξουμε. Σας ευχαριστούμε για αυτή την υπόδειξη και το προσέξαμε. Βέβαια το κλειδί για την αλλαγή είναι οι άνθρωποι, όπως πολύ συχνά ε, ε, αυτό συμβαίνει. Έχουμε ένα πρέσβη εξαιρετικό, έναν άνθρωπο που έχει αφιερωθεί ψυχή και σώματι στην αποκατάσταση της ΑΕΤΗΣ και έχουμε ε, ε, υπεύθυνη του ανθρωπιστικού μας προγράμματος μία ε, γυναίκα που πραγματικά είναι αφοσιωμένη και δουλεύουν μαζί και για να αποκαταστήσουν τις γειτονιές και για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από τις καταστροφές και για να υπάρξει παράλληλα και εκπαίδευση και υγεία και για να καταπολεμήσουν τη χολέρα. Είδα επιτόπου έξι προγράμματα που με εντυπωσίασαν και γύρισα έχοντας δει πολλά στην IT. για τους δωρητές υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να στυλιτεύσουμε, διότι ξεκινήσαμε με πολλά χρήματα, 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μια χώρα που δεν έχει θεσμούς που θα μπορούσαν να απορροφήσουν τόσα χρήματα και τρία χρόνια αργότερα ακόμη ε, χτίζονται αυτοί οι θεσμοί και δεν μπορούν να απορροφηθούν 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέτοιο περιβάλλον. Άρα δεν προχωρούν πολύ γρήγορα τα διάφορα προγράμματα. Αυτό οφείλεται στο ότι θέσαμε μη ρεαλιστικές προσδοκίες και ανησυχώ, διότι μπορούν οι δωρητέ να πούν «Α, βλέπεις, δεν προχωράνε τα προγράμματα, να μειώσουμε τη χρηματοδότηση». Αυτό θα ήταν τεράστιο λάθος. Γιατί η IT δεν είναι ένα τριετέ πρόγραμμα, είναι ένα τριακονταετέ πρόγραμμα, αν θέλουμε να έχουμε την δέουσα σοβαρότητα. Έτσι, έτσι Έχετε λοιπόν. δίκιο. Να, να συνεχίσουμε τον κύριο Γκέρεντς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και να συγχαρώ την Επίτροπο, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρουσία της σήμερα εδώ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, ούτε για την κατάσταση που μας περιγράψατε στο Μάλι, ούτε για την κατάσταση στη Συρία. Θα ήθελα παρόλα αυτά να σας πω ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο Μάλι για να επανέλθει η σταθερότητα ήταν τόσο ραγδαία που αναρωτιόμαστε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πού πήγαν οι τρομοκράτες, διώχτηκαν, Πού είναι όμως, εξαφανίστηκαν. Η απάντηση σαφώς είναι όχι. Μου θυμίζει κάτι που ήδη το γνωρίζουμε, μου θυμίζει την κατάσταση του Αφγανιστάν. Ραγδαίες εξελίξεις στρατιωτικές και κατόπιν επανεμφάνιση των τρομοκρατών με τρομερά προβλήματα επί χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι σήμερα η συνεργασία υπό την αιγίδα είτε των κρατών μελών είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύουν και το θέμα της ασφάλειάς τους θα πρέπει να το εγγυηθούν κάποιοι. Ποιοι θα το αναλάβουν αυτό από εδώ και πέρα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ενώ συμφωνώ απολύτως με τα πολύ επενετικά σχόλια όσον αφορά την εργασία που κάνει η διεύθυνσή σας στην Επιτροπή. Θα ήθελα να πω ότι εδώ γίνεται ένα τεστ, μία δοκιμή της α, ε, ε, αμεροληψίας της δράσης σας. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτές τις σειράξεις. Και αυτό ισχύει και για τη Συρία, αλλά όχι μόνο για τη Συρία. Και καταλαβαίνω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα τμήματα που συνεργάζονται για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνομιλούν και συνεργάζονται. Αλλά κάπου υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα χωρίς τέτοια προηγούμενη συνεργασία και εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την αμερόληπτη ε, δράση σας. Συμφωνούν όλοι με αυτή την προσέγγιση. Αυτή είναι η συμπληρωματική μου ερώτηση. Και τέλος, Η συζήτηση όσον αφορά το πολιετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο έχουν οδηγήσει σήμερα στην Ευρώπη σε μια κατάσταση που κινδυνεύουμε να μην μπορέσουμε να συλλέξουμε τους απαραίτητους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι η δική σας δράση δεν θα μπορέσει να υποστηριχθεί καθότι θα λείπουν σημαντικά κονδύλια. Πώς βλέπετε αυτές τις προοπτικές στο μέλλον. Είναι διατεθειμένα τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή δράση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ό,τι δηλαδή δεν δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμπληρωθεί από περισσότερες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο. Σας άκουσα με μεγάλη χαρά να λέτε ότι εσείς θα κάνετε ό,τι μπορείτε και όσον αφορά τους κοινοτικού πόρους, αλλά και για να πείσετε τα 27 κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε το πώς τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν τις δεσμεύσεις τους τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις κοινέ αρμοδιότητες που έχουν. Και δεν θα πρέπει εδώ κανείς να μην αναλάβει τις ευθύνες του. Και εδώ αναφέρομαι και στις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες που είναι ο έλεγχος, αλλά και μια πολιτική κινητοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ντέβα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μερικές φορές όταν ακούμε τι κάνει η Κομισιόν στο όνομα των ανθρώπων της ε, Ευρώπης, νιώθουμε περήφανοι για τη δουλειά που κάνει. Αυτά που μόλις ακούσαμε είναι πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Ως ε, Ευρωπαίοι ε, φορολογούμενοι βοηθήσαμε τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και που ε, είναι πιο ευάλωτοι και στο Μάλι και στη Σύρια. Επικροτώ και τη δουλειά της ΕΚΟ και της Κομισιόν. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά για να σώσετε ζωές, πιθανότητα των πιο ευάλωτων ανθρώπων ε, στον πλανήτη. Αλλά εάν εξετάσουμε ολιστικά τα θέματα αυτά και όχι από ανθρωπιστικής πλευράς, αναρωτιέμαι τι ακριβώς κάνουμε. Διότι... Στο Μάλι έχω την εντύπωση, όπως υπόθηκε, ότι θα ξεκινήσει ο ανταρτοπόλεμος ε, από τους ε, τζιχάντ. Έτσι θα έχουμε αστάθεια και θα εμποδιστεί η ε, επανεγκατάσταση των ανθρώπων, καθώς και ένα σταθερό κλίμα για την ανάπτυξη. Ποια είναι λοιπόν η απάντησή μας σε αυτές τις περιπτώσεις που οι αντάρτες αποσύρονται στην έρημο, ξαναχτυπάνε στις διάφορες περιοχές, θα έχουμε πιο πολλούς πρόσφυγες. Ποια είναι η λύση μας. Αυτό το είδαμε στο Αφγανιστάν. Εδώ και χρόνια στο Αφγανιστάν το βλέπουμε και με έναν απλό υπολογισμό έχουμε δαπανίσει 3.700 ευρώ ανά Αφγανό από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα. Θα γνωρίζετε ότι το ε, κατακεφαλήν ΑΕΠ ε, ε, στο Αφγανιστάν είναι 600 δολάρια, 500 ευρώ περίπου. Εφτά φορές το ποσό, έχουμε εξοδέψει το εφταπλάσιο ανα Αφγανό. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα εγκαταλείψουμε τη χώρα και θα την αφήσουμε στα χέρια των Ταλιμπάν. Γιατί πήγαμε εκεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε μια ολική κατανόηση του τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Δαπανίσαμε τεράστια ποσά στο Αφγανιστάν. Για ποιο σκοπό ακριβώς. Και τι θα πετύχουμε στο Μάλι αν δεν έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Φυσικά πρέπει στην ανθρωπιστική βοήθεια να κάνουμε αυτά που πρέπει, αλλά θα πρέπει και άλλοι να κάνουν τα απαραίτητα για να πετύχουμε ειρήνη. Και στη, Σύρια, και στη Συρία ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ε, Σύριους. Ε, και μίλησε η Κομισιόν για τα ποσά που θα χρησιμοποιηθούν για να παράσχουμε τροφή, νερό, ε, υπηρεσίες υγιεινής στη Συρία. Οι Άραβες τι κάνουν, Η Σαουδική Αραβία τι κάνει που είναι πλούσια, το Κατάρ τι κάνει, το Κουβέιτ τι κάνει, τι κάνουν όλοι αυτοί. Γιατί πάντα ο κακομοίρη Ευρωπαίος φορολογούμενος θα πρέπει να φέρει το μεγαλύτερο βάρος. Ε, θέλω απαντήσεις σε, αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόρτες Λάστα και κατόπιν θα απαντήσει η Επίτροπος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Γεωργίευα, και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δουλειά που έχετε κάνει. Όλοι νιώθουμε περήφανοι για τα όσα ακούσαμε. Για τα όσα κάνατε εσείς, μόλις γύρισα από την Κολομβία που έχει τον ε, δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων, 3 ε, με 4 εκατομμύρια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σχετικά με το Μάλι. Μιλήσατε για υπολογισμούς που γίνονται, την ανάγκη να έχουμε παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήταν ε, ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είδους ανταπόκριση είχατε στο θέμα αυτό. Είχατε παρατηρητές στο Μάλι που να εξετάζουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και στην περίπτωση της Συρίας θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Είπατε ότι η σύγκρουση εκεί πιθανότατα να κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα. Δεδομένου τούτου, έχουμε συναντήσεις συντονισμού και σχεδιασμού με ε, τον ΟΗΕ, με τον Ερυθρό Σταυρό, για να δούμε πώς μπορούμε να ενεργήσουμε από κοινού ώστε να μην έχουμε αύξηση από το 1 σε 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένων. Γίνεται συντονισμός όσον αφορά ε, τους καταβλισμούς προσφύγων κλπ. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Γεωργίεβα. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Ε, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Ε, στον κύριο Γκόνη, να πω ότι φυσικά συμφωνώ μαζί σα ότι ε, η στρατιωτική νίκη του μήνα αυτού ε, είναι σχετικά εύκολο ε, κομμάτι. Το να διατηρήσουμε την ασφάλεια μακροπρόθεσμα είναι πιο δύσκολο. Έχουμε εδώ μία περιοχή όπου εδώ και αρκετό καιρό έχουμε δει απαγωγές, ε, εμπόριο ναρκωτικών, πράγματα που έχουν ε, οδηγήσει σε υψηλά έσοδα για κάποιους ε, και έχουν ε, δώσει οικονομικούς πόρους στους εξτρεμιστές. Και αυτό δυσκολεύει πολύ το να αλλάξουμε την κατάσταση. Μου είπανε ιστορίες για 10.000 ευρώ για μεταφορά ναρκωτικών με ένα φορτηγό, για τον οδηγό του φορτηγού. Πώς θα κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, γεωργούς, πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε ε, όταν ε, πραγματοποιείται τέτοιο είδους εμπόριο. Όσο επιτυχής και να είναι η στρατιωτική παρέμβαση λοιπόν, δεν θα εκριζώσει τον εξτρεμισμό. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό να οικοδομήσουμε δυναμικό ε, ε, στρατού στο Μάλι, αστυνομίας ε, κλπ. Πρέπει όμως επίσης να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια μας. Τι είναι εφικτό. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό που είδαμε στην IT, όπου είχαμε τελείως μη ρεαλιστικές προσδοκίες δεν έχω να σας δώσω κάποια μαγική συνταγή. Το Μάλι είναι τυπική ε, περίπτωση. Έχουμε το ε, αρκετά χαμηλό κατόφλι της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας ε, έχουν αρκετή ανεκτικότητα ε, οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό λοιπόν ε, θέλουμε να παντρέψουμε αυτό με την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό είναι σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά το θέμα της αντικειμενικότητας είναι σημαντικό ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι μιλάμε για συνεχιζόμενη παρουσία σε ένα περιβάλλον που θα δει σημαντικές διακυμάνσεις ε, στο μέλλον για αρκετό χρονικό διάστημα. Στην Κομισιόν και στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, προοδεύουμε όσον αφορά τον καθορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων κατά τη συνεργασία μας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλαίσιο και έχουμε καθορίσει και τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο μέτωπο αυτό ε, με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Έχουμε δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση εντός της οποίας καθορίζουμε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της ανθρωπιστικής βοήθειας, πού συμμετέχουμε και πού όχι. Η ανάγκη για αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία θα διασφαλιστεί. Είμαι λοιπόν αισιόδοξη ότι περιπτώσεις όπως το Μάλι και η Συρία μας ε, διδάσκουν κάποια πράγματα περί πολιτικής, σχετικά με το πώς στο μέλλον μπορούμε να παράσουμε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, προφανώς ε, δεν είμαι σε θέση να πω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η Κομισιόν υπέβαλε την πρόταση, εμείς την βρίσκουμε καλή, τα κράτη-μέλη Ε, υπέβαλαν πρόταση, γίνονται διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, αλλά ελπίζω ότι στο τέλος θα δούμε αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, στον κόσμο τούτο με τους πολλούς κινδύνους. Και Τελικά πιστεύω ότι θα έχουμε ε, τις ε, απαραίτητες το, απαραίτητο δυναμικό και τους απαραίτητους πόρους στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μαζί μας τα κράτη-μέλη. Όταν η Κομισιόν στην περίπτωση μιας δύσκολης κρίσης Ε, θέλει να κάνει κάτι, τότε φέρει και όλο το βάρος της Ευρώπης μαζί της. Δεν ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να κάνουμε τη δουλειά των κρατών μελών. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη όσον αφορά το 0,7%. Δεν νομίζω ότι εξηγούμε επαρκώς στο κοινό μας γιατί είναι προς συμφέρον μας ε, να εμείνουμε στη δέσμευση αυτή. Για όλους μας νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί ακόμα και όταν έχουμε μέτρα λιτότητα στις πατρίδες μας θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε με τη δέσμευσή μας αυτή, διότι ε, εάν δεν το κάνουμε αυτό τότε θα έχουμε πολύ μικρότερη αγορά για τα προϊόντα μας και πολύ, μικρότερη, πολύ λιγότερη πολιτική σταθερότητα στην οποία να μπορούμε να ε, δραστηριοποιηθούμε. Θα ζητούσα από το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες του στο θέμα της ευελιξίας, διότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα εάν έχουμε την ευελιξία να προσαρμόζουμε τις αποφάσεις μας περί χρηματοδότησης. οι άλλοι μας συνάδελφοι είναι πολύ ε, πιο δεσμευμένοι, δεν μπορούν να ε, προσαρμόζουν τόσο πολύ τις αποφάσεις τους περί χρηματοδότησης όσο μπορούμε εμείς στον ανθρωπιστικό τομέα. Αν μου επιτρέπετε, ε, κύριε Γκέρενς, λέει η Πρόεδρος. δεν μπορείτε να πάρετε τη σειρά πριν από όλου του άλλου. Όχι, μόνο ένα σημείο ήθελα να αναφέρω, λέει ο κ. Γκέρεν. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, αδιαφορεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το δικό μας μήνυμα, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου από κοινού, θα είναι το να πούμε προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να διαφορεί το Συμβούλιο και για την ανθρωπιστική δράση και για την αναπτυξιακή δράση. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα πολύ σημαντικό που πλήττει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έρηδες μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω ότι αυτό αθετεί κάποιες υποχρεώσεις που έχουν δώσει στο παρελθόν. Το θέμα της ευελιξίας ε, μας το έχουν ε, αναφέρει και ο κύριος Βαναρόμπου και ο κύριος ε, Μπαρόζο. Εμείς πιστεύουμε ότι η ευελιξία δεν λύνει το πρόβλημα της απουσίας κονδυλίων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε ως μήνυμα από τη σημερινή μας συνεδρίαση. Προφανώς δεν θα διαφωνήσω με το γεγονός ότι δεν είναι προσυμφέρον της Ευρώπης να ξεχάσουμε ε, τις δεσμεύσεις που έχουμε κάνει απέναντι στο υπόλοιπο του κόσμου. Δεν μας βοηθάει αυτό. Ε, το βλέπω όταν ταξιδεύω. Ε, στοιχίζει όσον αφορά τη φήμη μας. Ε, και αυτό σημαίνει και απώλεια αξιοπιστίας. Ε, ωστόσο, όσον αφορά την ευελιξία, καλύτερο είναι να έχουμε περισσότερα χρήματα και περισσότερη ευελιξία, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά το θέμα αυτό. Και σας το λέω αυτό ως άνθρωπος που όλη μου τη ζωή ε, ασχολούμουν με του οικονομικούς πόρους. Όταν ε, ήρθα στην Κομισιόν από την ε, Παγκόσμια Τράπεζα, με εξέπληξε η, η ακαμψία που έχουμε κατά τη διαχείριση των πόρων μας και πόσο αυτό είναι η βάρος της επιρροής μας. Θα παρακαλούσα λοιπόν το Κοινοβούλιο να κάνει, προφανώς ότι είναι καλύτερο για την Ευρώπη. Να απαντήσω στον κύριο Ντέβα όσον αφορά την ολιστική προσέγγιση και το τι κάνουν οι αραβικές χώρες. Εμείς που ασχολούμαστε με την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του στρατιωτικού σχεδιασμού ή της πολιτικής δράσης. Δεν είναι δουλειά μας αυτό. Δουλειά μας όμως είναι να λέμε ότι εάν επιτρέψουμε γρήγορη απόσυρση των ε, στρατευμάτων σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ε, η δουλειά, ε, τότε σίγουρα επιδεινώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Όσον αφορά τι άλλε χώρε. το Κουβέιτ έδειξε πολύ ισχυρή παρουσία. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε 300 εκατομμύρια, επίση και το Κουβέιτ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα άλλα 300 εκατομμύρια. Έχουν υποσχεθεί λοιπόν να διαθέσουν ποσά και βλέπουμε να τηρούν τις υποσχέσεις τους. Τους επενώ λοιπόν για τις δεσμεύσει αυτές και μάλιστα το κλίμα στο ε, Κουβέιτ ήταν ε, ε, πολύ νυφάλιο. Εγώ νόμιζα ότι θα ακούγαμε πολιτικές ε, ομιλίες κλπ. Όχι, όλοι ήταν επικεντρωμένοι στην ανθρωπιστική κατάσταση επειδή ακριβώς είναι τόσο σοβαρή. Ε, ακόμα θα πρέπει να αναπτύξουμε μια κουλτούρα ε, διαφανούς λογοδοσίας ε, μεταξύ των, των χορηγών και μάλιστα καλό τον ΟΤΣΑ, τον Οργανισμό Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ, να εκπονήσει έκθεση σχετικά με το ποιος έχει τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στο Κουβέιτ. Επίσης, Ε, υπάρχει θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά έχει προεκτάσεις ε, που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε τις αρχές του Μάλι. Έχουμε αυξημένη παρουσία του ΟΗΕ, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ελπίζω λοιπόν ότι οι αρχές του Μάλι θα συμφωνήσουν σε μεγαλύτερη παρουσία παρατηρητών για τα, για ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, προς το παρόν ε, είναι σχετικά περιορισμένο το δυναμικό. Και όσον αφορά τον συντονισμό όσον αφορά τη Συρία, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με άλλους η ΕΚΟ, η δική μας υπηρεσία μαζί με την UNOSA και την Αραβική Λίγα, έχουμε δημιουργήσει το ε, Ανθρωπιστικό Φόρουμ για τη Συρία, το οποίο μάλιστα ε, θα συγκληθεί αύριο στην Γενέβη. Εφτά συναντήσεις είχε μέχρι στιγμής και εκεί συζητάμε ποιος θα κάνει τι, ποιες είναι οι ανάγκες, πόσο μεγάλο μέρος τους έχουμε καλύψει. Επίσης έχουμε επιτόπου συντονιστικές ε, συναντήσεις. Προσωπικό της ΕΚΟ συμμετέχει ενεργά κατά τον συντονισμό αυτών. Αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, διότι οι συνθήκες αλλάζουν. Και μάλιστα ο δύσκολο συντονισμό είναι αυτό με την αντιπολίτευση και με την κυβέρνηση, διότι οι συνθήκες ε, στι διαμάχε αλλάζουν κάθε μέρα. Μπορεί το πρωί να έχει κανεί πρόσβαση σε κάποια περιοχή και το απόγευμα ε, ο κόσμο να πυροβολεί τους, ε, ανθρώπου ανθρώπους που εργάζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο το κλίμα. Λοιπόν, τέσσερις ερωτήσεις και μαζί και οι απαντήσεις τους σε τέσσερα λεπτά, άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό το πολύ, κυρία Φροντνέρ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Για τη Συρία θέλω να μιλήσω στις ε, περιοχές των εξεγεθέντων. Εδώ νομίζω ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα και ο Ερυθρός Σταυρός ε, δεν ε, έχει εξίσου καλά αποτελέσματα όσο στις άλλες περιοχές. Δεν μπορούμε να δώσουμε άμεσα σε εξεγεθέντες και υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες. Ξέρουμε όμως ότι χρειάζονται περισσότερα και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για αυτούς που είναι ήδη παρόντες εκεί, για τους γιατρούς χωρίς σύνορα παραδείγματος χάρη. Τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει πιο ισορροπημένη η κατάσταση. Είμαι σίγουρη ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν θα έλεγα να δώσουμε βοήθεια άμεσα στους επαναστάτες, αλλά πρόβλημα υπάρχει. Κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω και εγώ τις αμφιβολίες του Σάχλα σχετικά με τις εξελίξεις στο Μάλι παρά την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού σήμερα που μας είπε ότι θα γίνουν οι εκλογές στις 31 Ιουλίου. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιο σενάριο όπως στο Αφγανιστάν, αλλά ίσως όπως στη Σομαλία. Και, εν περιπτώσει, μπορεί να έχουμε επιστροφή στο συνταγματικό δίκαιο, αλλά να παραμείνουν ε, οι επιθέσεις, στοχευμένες επιθέσεις. Ε, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, ακούσαμε σήμερα ότι υπάρχουν 400.000 πρόσφυγες σε άλλες χώρες έξω από το Μαλί και θα θέλαμε και θα ήθελαν στο Μάλι να επιστρέψουν για τις εκλογές στις 31 η Ιουλίου. Πώς θα γίνει η υποδοχή αυτών των προσφύγων, έχει προβλεφθεί κάτι, υπάρχει κάποια οργάνωση, θα παρεμβείτε κι εσείς σε αυτό Νομίζω ότι αυτό τίθεται ως ερώτημα. Κατά τα άλλα, το να κάνουμε τη χώρα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της ε, ε, είναι κάτι συζητήσιμο. Ξέρουμε ότι ε, η βοήθεια που δίνουμε για την ανάπτυξη δεν μπορεί να συμπιεστεί και είναι πολύ δύσκολο να τηρήσουμε αυτές τις υποχρεώσεις σε μια προσπάθεια σε μια περίοδο κρίσης. Ε, η βοήθεια για την ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμπιέσουμε. Συμφωνώ πολύ. Ο κύριος Μπέρμαν, θέλετε να λάβετε το λόγο για τη σύγκριση μεταξύ Αφγανιστάν και Μάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Μάλι είναι διπλάσιο σε μέγεθος με 15 εκατομμύρια πληθυσμό. Το Αφγανιστάν έχει 30 εκατομμύρια και τα 15 εκατομμύρια των κατοίκων του Μάλι δεν έχουν σύγκριση με τους Αφγανούς όσον αφορά το συντηρητισμό τους. Οι Αφγανοί υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των Ταλιμπάν, παρότι θέλουν σύνταγμα και θέλουν να ζήσουν σε διαφορετικό κόσμο από αυτόν που προτείνουν οι Ταλιμπάν, βρίσκονται πολύ κοντά τους κατά πλειοψηφία, πράγμα το οποίο δεν ισχύει στο Μάλι. Αντιθέτως, οι κάτοικοι στο Μάλι χαιρετίζουν την άφηξη των Γάλλων ε, γιατί θέλουν την επάνωδο της, του νόμου και της τάξης και της δημοκρατίας. Μπορεί να μην τα έχουν καταφέρει πολύ καλά, παρόλα αυτά ε, είναι αφοσιωμένοι σε αυτή, στο μέλλον τους ως δημοκρατία. Η καλλιέργεια του οποίου στο Αφγανιστάν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορούμε να ξεριζώσουμε, ενώ στο Μάλι δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα, δεν υπάρχει καλλιέργεια οπιούχων. Υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών, το οποίο διαφύρει ε, το λαό. Όντως είναι πρόβλημα, όπως ε, εξήγησε η Κρυσταλίνα Γεωργίευα. Και υπάρχει πρόβλημα διακίνηση ναρκωτικών και ε, διάβλων ναρκωτικών προς την Ευρώπη. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολη η συγκρίση μεταξύ Μάλι και Αφγανιστάν. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο. Κυρία Γεωργίευα. ξεκινώντας με την κυρία Μπρότνερ. Θέλω να πω ότι έδωσα κάποια παραδείγματα αυτών που κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτούς που βρίσκονται στις περιοχές που ελέγχονται από τους επαναστάτες και υποστήριξη από τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο ιδίω έχουν γίνει πάρα πολλά και παίξαμε και εμείς σημαντικό ρόλο επιμένοντας να χρηματοδοτηθούν τέτοιες δράσεις για να υποστηρίξουμε την παροχή βοήθειας ε, στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μέσω των φορέων που μπορούν να παρέχουν αυτή τη βοήθεια επιτόπου. Δεν θα αναφέρω ποιοι είναι αυτοί οι φορείς για να μην βάλουμε σε κίνδυνο τους εταίρους μας αλλά να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε κάθε δυνατό διάβλο για να φτάσει η βοήθεια στους ανθρώπους επιτόπου. Εγώ δεν θα κατηγορούσα τον Ερυθρό Σταυρό πάντως γιατί η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού πραγματικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Και αν δείτε το χάρτη, σε κάποιες περιοχές και σε αυτές που έχουν κόκκινα σημαδάκια, ε, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού μπορεί να παράσχει βοήθεια. Όσον αφορά την Ερυθρά ημισέλινο της Συρίας, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, διότι θεωρούνται κυβερνητικός φορέας. Και, και γι' αυτό στις περιοχές που ελέγχονται από τους επαναστάτες είναι πολύ δύσκολη η παροχή βοήθειας από την Ερυθρά ημισέλινο της Συρίας. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε με τον περισσότερους ε, ανθρώπους και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Χρησιμοποιούμε κάθε πιθανό διάβλο που θα μας βοηθούσε να φτάσει η βοήθεια στους ανθρώπους επιτόπου. Και είμαστε σε επαφή με την μονάδα βοήθειας και επισκέψεις έχουμε κάνει και έχουμε και συνεχή επαφή μαζί τους και είμαστε σε επαφή με όλους εκείνους που μπορούν να παράσχουν βοήθεια. Δεν έχουμε λοιπόν προκαταλήψεις με μία εξαίρεση. Δεν δίνουμε χρήματα απευθεία στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Ποτέ δεν δίνουμε βοήθεια κατά αυτόν τον άμεσο τρόπο. Ποτέ δεν το κάναμε και δεν θα το κάνουμε. Αλλά χρηματοδοτούμε τους εταίρους μας για να μπορέσουν να παράσουν βοήθεια. Είναι πολύ δαπανηρές οι δράσεις που έχουμε για να περάσουμε τις, γραμμές, τις εχθρικές γραμμές. Περιέγραψα προηγουμένως τις δράσεις που κάνουμε με αεροπλάνο που φτάνουν στη Λατάκια και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσει η βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. και να θυμάστε ότι για βοήθεια που έρχεται από άλλες πλευρές, όσον αφορά την Τουρκία ή και το Ιράκ, έχουν και εκείνοι κάποιους περιορισμούς στο τι θα εγκρίνουν. Και οι εγκρίσεις για ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι κάτι το τόσο εύκολο να, δοθεί, να δοθούν. Προσπαθούμε πάντως να φτάσει η βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. Μερικές φορές ε, δεν ε, τονίζουμε κάποιες δράσεις που κάνουμε, γιατί δεν γίνονται πάντα αυτές οι δράσεις με απόλυτη ασφάλεια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έδωσε βοήθεια σε περιοχές που ελέγχονται από τους επαναστάτες και αυτό μάλιστα ε, έλαβε δημοσιότητα έδωσαν βοήθεια σε ένα νοσοκομείο. Αυτό μαθεύτηκε και την επόμενη, το επόμενο βήμα ήταν ότι η κυβέρνηση βομβάρδισε το νοσοκομείο. Ε, η κρίση στη Συρία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πραγματικά χάνω τον ύπνο μου για αυτή την υπόθεση. Είναι πολύ δύσκολο περιβάλλον αυτό. Για την ερώτησή σας σχετικά με την υποχρέωση να επιστρέψουν οι πρόσφυγες. Αυτό δεν το κάνουμε ποτέ. Είναι μόνο ε, εκούσια η επιστροφή τους. Αν θέλουν να επιστρέψουν ε, στα σπίτια τους, επιστρέφουν. Και δεν συμφωνώ με το να πιέσουμε να γυρίσουν, να ψηφίσουν. Ε, συγγνώμη, λέει κυρία Ντεκάιζερ, παρανόηση υπήρξε εδώ. Θα είναι πολύ δαπανηρό εννοούσα το να επιστρέψουν. Οι οικειοθελώς θα επιστρέψουν, αλλά θα είναι πάρα πολύ δαπανηρό αυτό. Λοιπόν, ναι. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι το να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες στο βορρά ούτω ώστε να είναι οι συνθήκες εξίσου καλές ή και καλύτερες και αυτό να αποτελέσει μαγνήτη για τους πρόσφυγες ούτω ώστε να επανέλθουν. Δεν θέλουμε να ταξιδέψουν για να ψηφίσουν και να ξαναφύγουν. Πάντως όπως σας είπα και στην αρχή είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες στο Μάλι. Και συμφωνώ με τον κύριο Μπέρμαν ότι είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις του Μάλι και του Αφγανιστάν, όπως είναι διαφορετική και η Συρία από τη Λιβύη. Και κάθε φορά εξετάζουμε και τις ομοιότητες και τις διαφορές σε κάθε περίπτωση κρίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Γεωργίευα που ήρθατε στη συνεδρίασή μας και μας δώσατε τη δική σας εικόνα για τις κρίσεις αυτές που είναι διαφορετικές η μία από την άλλη. Η Επιτροπή Ανάπτυξης σας υποστηρίζει πλήρως τη δουλειά σας για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Σας υποστηρίζουμε και στην υπεράσπιση των ανθρωπιστικών αρχών έναντι όλων των πλευρών στις διενέξεις. Πάντοτε το κάνατε αυτό με μεγάλο πάθος αλλά και με διάβγεια και σας ευχόμαστε καλό κουράγιο στην επιδίωξη αυτών των ανθρωπιστικών στόχων. Και ελπίζουμε ότι στην επόμενη συνεδρίαση που θα σας έχουμε κοντά μας θα μας φέρετε και καλύτερες ειδήσει ή τουλάχιστον κάποιες θετικές εξελίξεις. Ευχαριστώ.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 Να συνεχίσουμε λοιπόν πριν φύγουν όλοι και μείνουμε μόνοι μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα άλλο ευαίσθητο θέμα από την ημερήσια διάταξή μας η κατάσταση της διατροφής και της γεωργίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως γνωρίζετε, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα κάθε χρόνο εκδίδει μία έκθεση με μία πλήρη εικόνα και υπάρχουν θέματα κέρια σημασία ε, για την ε, γεωργική ανάπτυξη και για την ασφάλεια των τροφίμων διεθνώ. Η τελευταία έκθεση με τον τίτλο «Επένδυση στη Γεωργία για ένα καλύτερο μέλλον» τονίζει τη σημασία τη επένδυσης στη Γεωργία και τονίζει και το ρόλο της ε, γεωργίας και των επενδύσεων εκεί ως μια στρατηγική από τις πλέον αποτελεσματικές για να μειώσουμε την ε, φτώχεια και την πείνα και για να προωθήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον κύριο Κώστα Σταμούλη που είναι Διευθυντής του Τμήματος ε, Οικονομίας Γεωργικής Ανάπτυξης του ΦΑΟ που θα μας παρουσιάσει τις βασικές γραμμές αυτής της έκθεσης και καλωσορίζουμε και την κυρία Στίνα και Ανέμα της Concord που θα λάβει το λόγο μετά την παρουσίαση του κυρίου Σταμούλη για να μας πει ποια είναι η θέση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα της ανάπτυξης. Κύριε Σταμούλη, έχετε το λόγο επί 20 λεπτά. Um, good afternoon. Thank you, Chair. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Κώστας Σταμούλης και είμαι διευθυντής ε, του τμήματος ε, αναπτυξιακής οικονομίας στη Γεωργία το τμήμα του ΦΑΟ στη Ρώμη και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία σήμερα να σας παρουσιάσω ε, την έκθεση για την επένδυση στη Γεωργία για ένα καλύτερο μέλλον. Το 2012 είναι η 65η επέτειος αυτής της έκθεσης ε, του ΦΑΟ που ε, ασχολείται με τα θέματα ασφάλειας τροφίμων ε, και φτώχειας. Και η φετινή έκθεση μιλά για το ρόλο των επενδύσεων στη γεωργία χάρη ενός καλύτερου μέλλοντος. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσιεύσεις για την κατάσταση των τροφίμων και τη γεωργία το 1947 και το 1949 συγκεκριμένα. Ορισμένα από τα θέματα τα οποία συζητούνταν τότε συζητούνται και το 2012. Στις εκθέσεις λέει του 1947 και του 1949. Και οι συστάσεις ε, σε μεγάλο βαθμό είναι παρόμοιες. Δηλαδή η καμπύλη μάθησης βλέπουμε ότι καμιά φορά δεν είναι όσο βαθιά θα θέλαμε να ήταν. Το κίνητρο του να γράψουμε μία έκθεση για τις επενδύσεις στη Γεωργία ήταν το ότι η Γεωργία είναι το επίκεντρο της προσοχής όλων μετά τις ε, κρίση στον τομέα των τροφίμων, ιδίω μετά την πρώτη τέτοια κρίση. Και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι τελικά η γεωργία έγινε τμήμα της αναπτυξιακής συζήτησης, όπως και θα όφιλε. Πέρα των βραχυπρόθεσμων ανησυχιών που δημιουργούν οι αυξήσει των τιμών το 2007-2008, ετέθησαν και πολλά ερωτήματα για το αν θα μπορέσει ο κόσμος ε, το 2050 να εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τις διατροφικές του ανάγκες. Όταν θα είναι τόσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός, θα μπορεί η γεωργία να παράσχει τα απαραίτητα τρόφιμα. δεν είναι δεδομένα πλέον τα, τα πράγματα και ίσως δεν έχουμε τα προνόμια που είχαμε στο παρελθόν. Εν τα στοιχεία που είδαμε δείχνουν ότι η γεωργία άρχισε να είναι επίκεντρο της προσοχής και αν δείτε ε, τις τάσεις ε, στην επίσημη παροχή βοήθειας για τη γεωργία, υπάρχουν ε, κάποιες τάσεις στα μέσα της δεκαετίας 2000-2010 που σχετίζονται με το περιβάλλον που ακολούθησε την κρίση των τιμών. Και είναι ενδιαφέρον αυτό, διότι το μερίδιο της επίσημης βοήθειας που πηγαίνει στη Γεωργία κατέρευσε μετά την εχμή το σημείο εχμής ε, του περίπου 17-18% της συνολικής επίσημης βοήθειας κατέρευσε στο περίπου 3% στα τέλη της δεκαετίας ε, του 90 και λίγο πριν ε, το 2000. Φαίνεται ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ακολούθησε την τάση των τιμών. Βλέπουμε και τις κυβερνητικές δαπάνες και τις επενδύσεις στη γεωργία που ακολουθούν την πτωτική τάση των τιμών. Δεν ξέρουμε αν αυξήθηκαν το 2007 απλώς διότι έχουμε ατελή στοιχεία για την κυβερνητική χρηματοδότηση. Και αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που θα ήθελα να μεταφέρω σήμερα, ότι η ποιότητα των δεδομένων δεν είναι επαρκής. Θα ήθελα να πω επίσης ότι το μερίδιο της γεωργίας μειώνεται ενώ αυξάνονται άλλοι τομείς όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία που είναι και αυτή κλειδί για την ανάπτυξη. Και αυτό μας κάνει ακόμη περισσότερο να αναλογιζόμαστε το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τους μειωμένους πόρους που διατίθεται για τη γεωργία. Επίσης, εδώ έχουμε την καμπύλη που αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Φαίνεται να υπάρχει μία ε, στροφή μετά τις αρχές του 2000. Η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική αν ε, εξετάσουμε τις τάσεις λεπτομερέστερα, διότι οι συνολικές άμεσες ξένες επενδύσεις για τις 27 χώρες ε, για τις οποίες έχουμε στοιχεία διπλασιάστηκαν από το 2007-2008, αλλά μόνο το 6% πήγαν στα τρόφιμα και τη γεωργία και μόνο 0,4% στον πρωτογενή τομέα. Τα περισσότερα κονδύλια πηγαίνουν στη μεταποιητική βιομηχανία του γεωργικού τομέα, άρα σίγουρα δεν βρίσκεται εκεί η λύση. Επίσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη γεωργία πήγαν στους τομείς επεξεργασίας, όπως είπαμε, στη Γεωργία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση προς τις ε, χώρες με το ανώτερο ή μέσο εισόδημα. Επομένως υπάρχουν ανησυχίες για το τι ισχύει για την ασφάλεια της διατροφής και για την περιβαλλοντική σταθερότητα βλέποντας ε, τις επενδύσεις που γίνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι σημαντική αυτή η διαφάνεια που σας δείχνω τώρα, διότι εδώ έχουμε τις πρωτογενείς επενδύσεις στη γεωργία. Δηλαδή αυτά τα οποία επενδύουν οι ίδιοι οι αγρότες στα αγροκτήματά τους και το γεωργικό τους κεφάλαιο. Φαίνεται ότι οι πρωτογενείς επενδύσεις στη γεωργία αυξάνονται, ίσως ως αποτέλεσμα εν μέρη ε, στην, της αύξησης των τιμών ε, από το 2003 και μετά. Αλλά πιο σημαντική είναι αυτή η διαφάνεια. Όταν μιλάμε για επενδύσεις στη γεωργία, μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις κυρίως, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ή κυβερνητικές δαπάνες. Και εγώ εξάλλου από εκεί ξεκίνησα σκοπίμως την παρουσίασή μου. Αλλά αν δείτε αυτά τα δεδομένα, βλέπετε ότι οι επενδύσεις, ε, οι ιδιωτικές επενδύσεις από τους ιδιοκτήτες είναι πολύ υψηλότερες ε, και από τις κυβερνητικές επενδύσεις και από την επίσημη ε, βοήθεια. Πενταπλάσια είναι η επένδυση των ίδιων των αγροτών από των κυβερνήσεων και της επίσημη αναπτυξιακή βοήθειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική η κινητοποίηση δημοσίων κονδυλίων για τη γεωργία, αλλά αν θέλουμε ε, να, υπάρξει, ε, να υπάρξουν σωστές επενδύσεις στη γεωργία και για την ενέργεια και για όλα τα προϊόντα, θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις από τους ίδιους τους ε, αγρότες. Να μην σας καθυστερήσω με λεπτομέρειες τώρα, σας ε, διαβεβαιώ όμως ότι ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους είναι σημαντική αυτή η έκθεση είναι όχι μόνο το ότι επικεντρώνεται στο τι, τι επενδύουν οι αγρότες και όχι τόσο στο τι κάνουν οι κυβερνήσεις, αλλά η έκθεση αυτή αναφέρει και το τι θα πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις. Λέμε τι θα πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις για να προωθήσουν τις επενδύσεις των ίδιων των αγροτών και για πρώτη φορά έχουμε μία βάση δεδομένων σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις στη Γεωργία. Και αυτό είναι κάτι νέο, δεν το είχαμε παλαιότερα. Ίσως ε, και γι' αυτό ε, δεν έχουν ε, γίνει οι αναλύσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Αυτή είναι η εικόνα των επενδύσεων στη Γεωργία. Θα με ρωτήσετε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει διότι οι αυξήσει του αγροτικού κεφαλαιακού εξοπλισμού είναι αυτό το οποίο αξιοποιεί περισσότερο, δίνει μεγαλύτερη αξία ε, στην αγροτική εργασία. Δηλαδή, αν θέλουμε να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε την απόδοση στη γεωργία για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και ε, θα πρέπει να, να δώσουμε στους ε, αγρότες τη δυνατότητα να επενδύσουν στη γεωργία. Η εικόνα αυτή σας δείχνει πώς οι γεωργικές κεφαλαιακές ε, ο γεωργικός κεφαλαιακός εξοπλισμός αναεργαζόμενο φαίνεται ότι αυξάνεται. Και σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε, ε, βλέπουμε τον ε, γεωργικό κεφαλαιακό εξοπλισμό ανααγρότη και αυτό καταπολεμά την, ε, τον αριθμό των υποδιατρεφόμενων. Δηλαδή, από τις χώρες που φαίνεται ότι θα καλύψουν τους στόχους της χιλιετίας για την καταπολέμηση της πείνας, αυξάνεται κατά 7% κατέτος ο ρυθμός αυτών που στους οποίους καταπολεμάται η, η πείνα. Όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια είναι συνολικά και θα μπορούσε κανείς να θέσει το ερώτημα του τι γίνεται αν δούμε πιο αναλυτικά τα δεδομένα. Αλλά η συνολική εικόνα δείχνει ότι καταπολεμάται η πείνα στο συνολικό πληθυσμό και αυτό οφείλεται στις επενδύσεις ε, στη γεωργία. Και αν δούμε ε, την αρχή της περίοδου για την υποσαχάρια Αφρική και για την ε, Νότια Ασία βλέπουμε ότι αυξάνεται το μερίδιό τους, αλλά παρουσιάζεται και μια αρνητική τάση στην, στις επενδύσεις σε αγροτικό κεφαλαιακό εξοπλισμό αναεργαζόμενο. Αυξήθηκε λοιπόν η πείνα διότι μειώθηκαν οι επενδύσεις. Στην υποσαχάριο Αφρική οι γεωργικές επενδύσεις είναι θετικές, 1,5% κατ' έτος. Όμως, είναι πολύ μεγαλύτερε οι αυξήσει στο εργατικό δυναμικό στη Γεωργία, αλλά υπάρχει αρνητική ανάπτυξη. Και θα πρέπει να αυξηθεί ο γεωργικός κεφαλαιακός εξοπλισμός, γιατί αυτό είναι το σημείο κλειδί για την καταπολέμηση της πείνας. Νομίζω ότι σας έχω δώσει τώρα μια ξεκάθαρη εικόνα. Και αφού ε, διαπιστώσαμε ότι οι ίδιοι οι γεωργοί είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν επενδύσεις, για, γιατί αυτό είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της πείνας, πρέπει να δούμε τι άλλο σημαίνει αυτό. Ας ε, δούμε κάποια στοιχεία πέραν των τιμών. Το ένα είναι η διακυβέρνηση. Βλέπουμε ότι το συνολικό επενδυτικό κλίμα Και εδώ χρησιμοποιούμε ε, τους ε, δίκ, ε, το δίκτυ του κράτους δικαίου στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος και του επενδυτικού κλίματος. Και βέβαια αυτό είναι κάτι που πηγαίνει πέρα από τη γεωργία. Βλέπετε ότι υπάρχει ίδια συσχέτιση όπως και με άλλους δείκτες, όπως είναι ο πολιτικός κίνδυνος, η διαφθορά, ο ευάλωτος χαρακτήρας κλπ οι συνολικοί στόχοι μας δείχνουν καλύτερη διακυβέρνηση και ε, καλύτερες, ε, μεγαλύτερες επενδύσεις στη γεωργία. Αν δούμε το, τη συνολική διακυβέρνηση και ε, το συνολικό περιβάλλον, είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι πλήρης η εικόνα, γιατί πρέπει να δούμε τους κυβερνητικούς φορείς που έχουν σχέση με τη γεωργία και με τις επενδύσεις από τους ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων και αυτά να τα συνδέσουμε με τη σταθερότητα όσον αφορά την καλλιεργήσιμη γη. Εμείς πιστεύουμε ότι κινούμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταρχήν, το Μάιο του 2012 η Επιτροπή για την Παγκόσμια Επιστηστική Ασφάλεια ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατοχή γης στο πλαίσιο της εθνικής ε, διατροφικής ασφάλειας. Και αυτό είναι τεράστιο βήμα μπροστά. Αυτές οι εκούσιες κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν από 108 ε, κυβερνήσεις ε, και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τον ιδιωτικό τομέα, από ερευνητικά ιδρύματα για τη γεωργία. Άρα είναι τεράστια η πολιτι... Ε, τεράστιος ο πολιτικός αντίκτυπος. Δεν είναι δεσμευτικά, γιατί κανείς δεν δεσμεύεται να ακολουθήσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και μόνο ότι ε, υπέγραψαν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές δημιουργεί μια ηθική δέσμευση. Μια άλλη πολιτική διαδικασία που έχει σχέση με τη διακυβέρνηση στη Γεωργία είναι η διαδικασία της έγκρισης ε, των αρχών της υπεύθυνη γεωργίας. Στην τρέχουσα εκδοχή τους ε, είναι υπό την αιγίδα της Επιτροπής ε, Παγκόσμιας Επιστηστικής Ασφάλειας και ο στόχος τους είναι να υπάρξει ευρεία πολιτική συνένεση από όλους τους εμπλεκόμενους, από τις κυβερνήσεις, από τον ιδιωτικό τομέα, από την κοινωνία των πολιτών κλπ για να καταλήξουν σε κάποιες αρχές κοινά συμπεφωνημένες, ε, ώστε να δίδεται καθοδήγηση προς τις κυβερνήσεις, προς τον ιδιωτικό τομέα, προς τους επενδυτές, αν θέλετε, ούτως ώστε να γίνονται οι σωστές επενδύσεις που θα υποστηρίζουν την επισητιστική ασφάλεια, θα σέβονται το περιβάλλον, θα αποφεύγουν την περιθωριοποίηση των μικρών αγροτών κλπ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία και είμαι βέβαιος ότι αν δεν το έχετε ακούσει σύντομα θα φτάσει και στα αυτιά σας γιατί θα αποτελέσει ένα νέο τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι μεγάλες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είτε με εγχώρια κεφάλαια, είτε με ξένα κεφάλαια. Σε δύο χρόνια θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και τον Οκτώβριο του 2014 η Επιτροπή για τη Διεθνή Επιστηστική Ασφάλεια θα χρειαστεί να εγκρίνει αυτές τις οικειοθελείς κατευθυντήριες γραμμές. Πιστεύουμε ότι το περιβάλλον πολιτικής για τις αναπτυσσόμενες χώρες έχει βελτιωθεί όσον αφορά τις τιμές. Και η ανάλυση μας δείχνει ότι η γεωργία σε σχέση με άλλους τομείς έχει καλύτερες τιμές από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Το παγκόσμιο περιβάλλον όσον αφορά τις τρευλώσεις των τιμών έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν κατά αυτόν τον τρόπο τα κίνητρα όσον αφορά τις τιμές για να μπορέσουν να επενδύουν οι αγρότες. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα περάσω στο εξή. Όπως είπα και προηγουμένως, η έκθεση αυτή δεν μειώνει το θεμελιώδη ρόλο που παίζουν οι κυβερνήσεις και η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, διότι αυτοί αποτελούν καταλύτες για την πρόθεση της, των επενδύσεων των αγροτών. Είδαμε ότι οι επενδύσεις από τις κυβερνήσεις σε βασικά αγαθά. Εδώ το παράδειγμα που βλέπετε αφορά την Κίνα, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στην έκθεση. Έχουν ως αποτέλεσμα και τη μείωση της φτώχειας και κέρδη για τους αγρότες. Δεν υπάρχει λοιπόν αντίφαση μεταξύ των δύο. Παράλληλα, η απόκτηση ιδιωτικών αγαθών μέσω, μέσω επιδοτήσεων δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό μέσο. Άρα, τα βασικά μας μηνύματα. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι θέλετε να τελειώνω την παρέμβασή μου. Η επενδύση στη γεωργία είναι μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση της πείνας. Οι αγρότες είναι αυτοί που παίζουν βασικό ρόλο και πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς παράγοντες στη στρατηγική μας και θα πρέπει να διαμορφώσουμε την πολιτική κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επενδύουν οι ίδιοι αγρότες. Επίσης είναι αποτελεσματικό, είναι απαραίτητο, ε, αλλά όχι επαρκές, ένα θετικό επενδυτικό κλίμα. Θα πρέπει να ε, δείξουμε μεγάλη προσοχή για τους μικρούς αγρότες που χρειάζονται ειδική βοήθεια και οι μεγάλες επενδύσεις, οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας χρειάζονται ειδική ε, προσοχή. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εστιάσουν στα δημόσια αγαθά με υψηλή απόδοση και ε, χρειάζομαστε μια πολύ καλύτερη βάση τεκμηρίωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξεπεράσατε το χρόνο σας και αυτό είναι εις βάρος των υπόλοιπων ομιλητών. Γι' αυτό προσπαθώ να είμαι πιο αυστηρή. Η επόμενη ομιλήτρια για 7 λεπτά έχει το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λέγομαι στην Εκούνεμα και εργάζομαι για την ΕΚΟ, μια οργάνωση μη κυβερνητική και σας ομιλώ εξ ονόματος της πλατφόρμας Concord, στην οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τις σκέψεις μας όσον αφορά τις απαραίτητες επενδύσεις για να υπάρξει περισσότερη επένδυση στον τομέα των ε, ειδών διατροφής και της επιστημιστικής βοήθειας. Δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας, αλλά επενδύσεως για να μπορέσουμε να παρέχουμε σε όλους την απαραίτητη διατροφή. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σταθερότητα στι επενδύσει στη γεωργία και να δώσουμε τα μέσα σε όλου όσου το χρειάζονται να μπορέσουν να παράγουν οι ίδιοι τα ίδια αυτά αντιδοφή. Παίρνουμε σαν σημείο κίνηση του γεωργούς, τους αγρότες και θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορέσουμε να καλύψουμε τι ανάγκε των ίδιων των γεωργών για επενδύσει, για να μπορέσουν να παρέχουν επιστημιστική ασφάλεια για του ίδιου και για τι οικογένειε του, σε μικρέ γεωργικέ να στηρίξουμε τις επιλογές τους, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να χρησιμοποιούν λιγότερο δαπανηρές τεχνικές και να καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών και περιφερειακών αγορών. Οι ίδιες οι ανάγκες των ε, γεωργών, πώς αυτές θα καλυφθούν σε λογικές τιμές. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη καταρχήν έτσι ώστε να στηρίξει αυτούς τους στόχους και να βοηθήσει τους αγρότες να επενδύσουν στις ίδιες τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Ποια είναι η πολιτική στην Ευρώπη, η κοινή αγροτική πολιτική καθώς και η διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα στην ε, Ρώμη όσον αφορά τι απαραίτητε επενδύσει στον τομέα των διατροφή, τη επιστική βοήθεια και τη συνοχή αυτή τη πολιτική κάτι το οποίο σαφώ θα πρέπει να ενσωματωθεί και σε όλους τους άλλους ε, στόχου. Η και ασφάλεια. Πρόκειται για ένα έγγραφο πολυσέλιδο το οποίο έχει προετοιμαστεί και δημοσιευθεί το 2010. Παρ' όλα αυτά, η υλοποίηση κανονικά θα πρέπει να στηρίζεται σε τρία σημεία, στην επιστημιστική ασφάλεια, καθώς και την ανάγκη να καλυφθούν οι ανάγκες για επισητιστική βοήθεια και να ενδυναμωθούν οι μικρή παραγωγή, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα ο ρόλος των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση αυτού του προγράμματος και να παίξουμε έναν ε, διευθυντικό ρόλο, πιλωτικό ρόλο. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της βιοπικιλότητας και η βοήθεια στους μικρούς παραγωγούς έτσι ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση στις τοπικές περιφερειακές αγορές. Επίσης, καλύτερος συντονισμός με τα προγράμματα επενδύσεων των κρατών και των περιφερειών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να λάβουμε υπόψη μας και τα διάφορα προγράμματα επιστημιστικής βοήθειας και υποστήριξης. Γι' αυτό και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει την υλοποίηση αυτών των στόχων και να ενσωματώσει όλους αυτούς τους στόχους στην υλοποίηση. Πρέπει επίσης να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το ότι η υλοποίηση αυτή θα πρέπει να περιέχει και την, τον τρόπο να υπάρξει συνοχή, να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και να δίνεται αναφορά από μέρους αυτών που καλούνται να υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Η Concord έχει ήδη κάνει δηλώσεις τα δύο προηγούμενα χρόνια για να μπορέσει η πολιτική αυτή να λάβει υπόψη τους περιβαλλοντολογικούς στόχους και για μας μια πολύ σημαντική πτυχή της απαραίτητης ε, μεταρρύθμισης είναι ε, η παραγωγή που αφορά τις ε, ζωοτροφές και συγκεκριμένα η καλλιέργεια σόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα και θα σας το αφήσουμε εξάλλου στην αίθουσα που παρουσιάζει τους στόχους αυτού του προγράμματος. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε για την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα στην Ολομέλεια το Μάρτιο να συμπεριλάβετε διάφορες ε, τροπολογίες που να λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις προτάσεις αλλά και τα πρωτεϊνούχα όπως παραδείγματος χάρη τη σόγια και το καλαμπόκι. Ξέρουμε ότι υπάρχει επεξεργασία των προτάσεων αυτών και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και σας παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψη σας αυτές τις προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξει συνοχή στην πολιτική η οποία θα προταθεί από εσάς. Από τον συνάδελφο από την ΕΦΑΟ ακούσαμε τις προτάσεις ενός ανεξάρτητου δημοκρατικού οργανισμού για το θέμα της επιστημικής ασφάλειας, της διατροφικής ασφάλειας και θεωρούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πολιτική συζήτηση που λαμβάνει η χώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλαβαν χώρα διαβουλεύσεις και στη διαδικασία αυτή θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει συνοχή με την γενικότερη πολιτική της όσον αφορά τα ιδιοτροφίες και την επιστημιστική ασφάλεια. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την προαιρετική εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να λάβετε υπόψη σας αυτές τις διαβουλεύσεις πριν υιοθετήσετε την ε, ευρωπαϊκή θέση στηρίζοντας ε, τις μικρές ε, εκμεταλλεύσεις, τους μικρούς γεωργούς. Σας ζητούμε επίσης να αναλύσετε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διαδικασίες και εκτός της ε, διαδικασίας που συζητούμε σήμερα εδώ και σε άλλα πλαίσια. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να ε, προετοιμαστεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά την διατροφή. Δεν μπορεί να υπάρξει επιστηστική ασφάλεια χωρίς ε, ασφάλεια των ειδών διατροφής. Και θα θέλαμε εδώ να λάβουμε υπόψη μας τους συνδέσμους που υπάρχουν μεταξύ της γεωργικής παραγωγής, της επισητιστικής ασφάλειας, της ασφάλειας των ειδών διατροφής και να ληφθούν μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την ασφάλεια της επισητιστικής βοήθειας, των ειδών διατροφής, κάτι που θα είναι σαφώς προς όφελος των μικροκαλλιεργητών, των μικροπαραγωγών, κάτι που έχει συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη δήλωσή της. Σας ζητούμε λοιπόν να λάβετε υπόψη σας και να αναλάβετε το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων στην προετοιμασία την, ε, των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να φέρω, ξέρετε πολύ καλά ότι χρειάζεται συνοχή για την ε, προετοιμασία της ε, πολιτικής σας στον τομέα της επιστημιστικής ασφάλειας. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ των τομέων έτσι ώστε να φτάσουμε σε πραγματική ασφάλεια των ειδών διατροφής. Γι' αυτό και σας ζητούμε να συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας από άλλες επιτροπές όπως την Επιτροπή Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη η συνοχή όλων των μέτρων που καλείστε να υιοθετήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Πρόεδρος, ο κύριος Γκέρεντς είναι ο πρώτος που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας έκαναν. Θα ήθελα να πω στον εκπρόσωπο της ΦΑΟ ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω κάποιον να λέει με τέτοια σαφήνεια ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των τιμών υψηλών τιμών ή πιο υψηλών τιμών και των κινήτρων των γεωργών προς παραγωγή. Είναι τόσο αυτονόητο που έπρεπε να το πούμε παρόλα αυτά. Δηλαδή, από εδώ και πέρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια πολιτική καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Αν είναι σημαντική η επίπτωση των τιμών, θα σας πω ότι οι χαμηλές τιμές είναι κάτι που οδηγούν κάποιους ε, παραγωγούς στην εγκατάλειψη των καλλιεργειών. Και αυτό ισχύει και για την περιοχή του Σεχέλ. Σήμερα οι τιμές των δημητριακών είναι υψηλές και ο παραγωγός σε αυτή την περιοχή κερδίζει ένα δολάριο την ημέρα. Πριν από 10 χρόνια οι τιμές ήταν τέτοιες που του απέφεραν ένα κέρδος μισό δολάριο την ημέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επίπτωση των τιμών είναι καθοριστική. Σήμερα μιλάμε για έναν οικονομικό φιλελευθερισμό, μια απελευθέρωση και αυτό μας οδηγεί σε τιμές που δεν καλύπτουν πάντα τις ανάγκες των ε, πιο αδύνατων. Αυτό βεβαίως μας οδηγεί στο ερώτημα αν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε προστατευμένες αγορές. Και θα σας υπενθυμίσω ότι ο Εντιά που γνωρίζει τα γεωργικά θέματα, μίλησε για την διάσωση όλων των γεωργικών καλλιεργιών μια προστασία που δεν θα πρέπει να περιορίζεται παραδείγματος χάρη μόνο στην περιοχή του Σαχέλ αλλά παντού στον κόσμο καθότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια ταυτόχρονη δράση προστασίας των γεωργικών καλλιεργιών. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, του ΦΑΟ και της Κονκόρντ που ακούσαμε σήμερα. Στο παρελθόν, ε, στην Επιτροπή Επισητιστικής Ασφάλειας, ε, συζητήσαμε το θέμα των ε, αγροτικών συνεταιρισμών και θα ήθελα να ακούσουμε περισσότερα για τις δυνατότητες των συνεταιρισμών αυτών και αν μπορούν να αποτελέσουν ε, λύσεις στο πρόβλημα της ε, παροχής τροφίμων. Όσον αφορά την κατανομή των εκτάσεων, νομίζω ότι απομένουν πολλά να γίνουν, διότι είναι θέμα που συνδέεται άμεσα με αυτό που ανέφερε ο κύριος Γκέρενς, την, την μονοκαλλιέργεια, την καλλιέργεια μιας, ε, ενός είδους που έχει περισσότερα οικονομικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, όπου έχουμε πιο βιώσιμη γεωργία. Και επίσης κάτι που βλέπουμε να λείπει συχνά είναι η υποδομή για τη διάθεση των προϊόντων. Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Γεωργός όταν θέλει να απολύσει τις καλλιεργίες του. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Είναι προφανές ότι Ε, οι συλλογισμοί των μελών ε, του Κοινοβουλίου είναι παρόμοιοι με τους δικούς σας. Ε, πρόσεξα επίσης το διάγραμμά σας που δείχνει την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Αυτή η τάση μπορεί να είναι θετική για τους παραγωγούς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω στις τάσεις αυτές. Ε, εγώ γενικά στηρίζω τις τάσεις αυτές, διότι πιστεύω ότι τα, ε, τα τρόφιμα είναι υπερβολικά φθηνά. Οι περισσότεροι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά τις τιμές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, μπορείτε να μας πείτε τι ποσοστό της τιμής καταλήγει στον παραγωγό και τι ποσοστό χάνεται στα τούνελ, στο, στους ε, ενδιάμεσους, ε, στους μεταπολιτές, ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Ο Λεωνάρ Μηδία από την Επιτροπή. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θέλαμε να επικροτήσουμε τη δημοσιοποίηση της έκθεσης αυτής. Ε, μάλιστα, ήμασταν παρόντες κατά την παρουσίασή της ε, τον Δεκέμβριο ε, στη Ρώμη. Συμφωνούμε και με την έκκληση για δράση και όσον αφορά τις επενδύσεις. Συμφωνούμε και γενικά με τις με τους συλλογισμούς που παρουσίασε ο κύριος Σταμούλης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις συζητήσεις σχετικά με την επιστημιστική ασφάλεια, στην Επιτροπή για την Επιστημιστική Ασφάλεια και ε, σε διάφορες διαδικασίες. Για παράδειγμα, στο σχέδιο δράσης ε, του G, των G20 ε, που συμφωνήθηκε κατά το 2010 και 2011 από τους αρμόδιους υπουργούς. Εδώ παρακολουθούμε τις δραστηριότητες που ξεκίνησε η Γαλλική Προεδρία και που συνεχίζει η Μεξικανική Προεδρία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επενδύσεις μικρών εκμεταλλεύσεων και τις συμπράξει ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. και φέτος ε, θα συνεχίσει η επικέντρωση στην παραγωγικότητα και την ε, σωστή διαχείριση. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το θέμα της διακυβέρνησης ε, των γεών και της κατανομής των εκτάσεων, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Γι' αυτό επικροτούμε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αρμόδια διαχείριση των γεών. Ε, κατευθυντήριες γραμμές υιοθετήθηκαν πέρσι τον Μάιο και ε, ε, δεσμευόμαστε να συμμετάσχουμε στην πραγματοποίησή τους. Επίσης, συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Σταμούλη να υπάρξει ένα εθελοντικό πλαίσιο σχετικά με τις διοργικές επενδύσεις. Χρειάζεται ένα τέτοιο πλαίσιο για να καθοδηγεί τους επενδυτές της χώρες υποδοχής και τους ε, παραγωγούς. Θέλουμε μια γεωργία που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και του φυσικούς πόρους. Επίσης θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση ε, των, ε, της απόκτησης εκτάσεων μεγάλη κλίμακας. Τον Απρίλιο οργανώνεται εργαστήριο, κυρίως για να εξεταστεί τι γίνεται όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις στην υποσαχάρια Αφρική και για να αναλύσουμε πώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η αφρικανική ε, γεωργία σχετίζονται μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός ε, τομέας ε, μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες για να αυξήσουν την επιστημιστική ασφάλεια. Συμφωνούμε επίσης με την έκθεση ότι ε, θα πρέπει να ευαισθητοποιούν οι γεωργοί και ε, συμφωνούμε με την υποστήριξη των ε, συνεταιρισμών. Οι γεωργοί θα πρέπει να νιώθουν ότι είναι δική τους η διαδικασία μεταρρύθμισης και το Αφρικανικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης βλέπει επικριτικά τις μεγάλες τις τις ε, πιο μεγάλες επενδύσεις, τις παρασκευές επενδύσεις ε, και καθότι ε, έχουμε τη δεκαετία της, την δέκατη επέτειο της δήλωσης του Μαπούτου, της διακήρυξης του Μαπούτο, επικροτούμε τις αλλαγές στην Αφρική αλλά και σε μέρη της Ασίας η διαδικασία αυτή που θα οδηγήσει του χρόνου στο ε, έτος οικογενειακής γεωργίας. Ε, στόχο έχουμε να εντοπίσουμε τα κενά που υπάρχουν και θέλουμε να υπάρξει διεθνής συντονισμός μεταξύ των χορηγών. Τέλος, οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, θα ε, πρέπει να ε, θέσουν τις γεωργικές πολιτικές στο, πλαίσιο, στο γενικό πλαίσιο της ανάπτυξης για να στηρίξουν τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Θέλουμε να συνεχιστεί ο διάλογος με τις ε, περιφερειακές ε, κοινότητες ε, στην Αφρική, ώστε να διαπιστώσουμε πού μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η υποστήριξή μας. Θέλουμε ένα ισχυρό διαθεσμικό πλαίσιο για να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και για να δημιουργήσουμε συνέργειες. Πιστεύουμε ότι ο ΦΑΟ μαζί με την ΙΦΑΤ και άλλες διεθνείς οργανώσεις μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο. Ε, σαφώς πρόκειται για ε, σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία. Ε, να μιλήσω και για την πολιτική συνοχή. Όλες οι υπηρεσίες της Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί το, την πρόοδο στον τομέα αυτών στις διάφορες πολιτικές. Και θα δείτε επικαιροποιημένη έκθεση το 2013 που θα περιγράφει την πρόοδο στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σταμούλη, έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου δίνουν τη δυνατότητα να αναφερθώ σε κάποια σημεία που δεν πρόλαβα να τα αναφέρω στην παρουσίασή μου. Καταρχήν, η πρώτη και η τελευταία ερώτηση έχουν άμεση σχέση. Οι τιμές. Όταν μειώνονται οι τιμές, καθότι υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή στην γεωργία και μεγαλύτερη στήριξη, αν θέλετε, της γεωργίας. Όταν αυξάνεται η παραγωγικότητα, βλέπουμε τους γεωργούς στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες να βλέπουν μόνο ότι μειώνονται οι τιμές. Και κάποιες άλλες χώρες να ξεκινούν έναν ανταγωνισμό, κάτι που οδήγησε τις τιμές σε περαιτέρω πτώση. Επίσης, οι διαφορές στις τιμές στο εσωτερικό μιας χώρας, παραδείγματος χάρη, κάτι που εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Πρώτον, έλλειψη υποδομών, προβλήματα στις τοπικές αγορές. Δεύτερον, το θέμα που αναφέρεται που είναι η ενδιάμεση. Πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού σε κάποιες αγορές και υπάρχουν άτομα ισχυρά που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στη διευθέτηση αυτών των αγορών. Τρίτον, υπάρχουν και τα εσωτερικά προβλήματα κάποιων χωρών που όσον αφορά τη φορολογία, όσον αφορά την επιδότηση κάποιων καλλιεργιών οδηγούν σε κάποια αποτελέσματα τα οποία έχουν αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Ένα λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις τιμές στο εσωτερικό μιας χώρας στις ίδια επίπεδα με τα ισχύοντα στις περιοχές κοντά στα σύνορα και όταν μιλάμε για αύξηση τιμών, βλέπουμε ότι η αύξηση τιμών ξεκίνησε το 2003 και κάποιοι από τους γεωργούς της αναπτυσσόμενης χώρας επωφελήθηκαν από αυτό. Ας πάρουμε το χάρη κάποια από τα οπροκυπευτικά ξεκίνησε μια παραγωγή και εδώ αν κοιτάξετε παραδείγματος χάρη στην εικόνα αυτή ότι σε κάποιες περιοχές δεν υπήρξε βελτίωση της παραγωγικότητας. Δεν υπήρξε γιατί δεν υπήρχαν επενδύσεις. Αυξάνονται λοιπόν οι τιμές και την ίδια ώρα υπάρχει η σημαντική αύξηση των τιμών που ακολουθείται από διακυμάνσεις πολύ έντονες, κάτι που χαρακτηρίζει τις αγορές μετά το 2007. Αυτές οι διακυμάνσεις αυτές οι αβεβαιότητες, η ραγδαία αύξηση των τιμών αλλά και οι διακυμάνσεις οι πολύ σημαντικές οδηγούν στην διαπίστωση ότι οι γεωργοί δεν έχουν τα εργαλεία και τη δυνατότητα να σταθεροποιήσουν τις αγορές με πιο σταθερή παραγωγή, παραδείγματο χάρη. Κοιτάξτε τι έγινε παραδείγματο χάρη στην εγκατάλειψη κάποιων ε, καλλιεργειών ε, Προ όφελο άλλων, όπως παραδείγματο χάρη με το καλαμπόκι. Βλέπουμε κάτι που επίσης οδηγήθηκε καταρχήν από τις διακυμένσεις στι τιμέ. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι βεβαίως ε, φαινόμενα που πλήττουν τον καταναλωτή της, ε, στις αναπτυσσόμενες αυτές χώρες και δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις ανησυχίες των αναπτυσσόμενων χωρών και των πιο ευάλωτων ε, καταναλωτών στις χώρες αυτές. Η αύξηση της παραγωγικότητας για λόγους περιβαλλοντολογικούς, αλλά και για άλλους λόγους που δεν οδηγούν ε, αυτόματα σε μεγάλη αύξηση των τιμών. Αυτό προσπαθούμε να πούμε σε αυτή την έκθεση. Πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε μια πιο σταθερή ε, παραγωγή με την τήρηση κάποιων στόχων. Κάνατε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και θα σας απαντήσω ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική συνταγή που να λειτουργεί για όλες τις καλλιέργειες. Σε κάποιες περιπτώσεις η διαφοροποίηση είναι πολύ θετικό γιατί μοιράζεται ο κίνδυνος με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι επιλέγουν μόνο καλλιέργεια γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερα κίνητρα που τους προσελκύουν. Δεν πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να είμαστε υπέρ της μίας ή της άλλης επιλογής. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αύξηση της παραγωγικότητας για να καλυφθούν οι ανάγκες, οι ανάγκες παντού στον κόσμο και συμφωνώ ότι πολλές φορές για μας είναι πολύ χαμηλές οι τιμές και καταστρέφουμε ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής γιατί, γιατί είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Αλλά για μας, για μας είναι πολύ χαμηλές οι τιμές γιατί ξοδεύουμε, δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του προπολογισμού μας στην διατροφή. Καταλαβαίνετε ότι για άλλες περιοχές του κόσμου η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Υποδομές, βεβαίως, συμφωνώ και ένα τμήμα αυτής της έκθεσης αναφέρεται στο σημείο αυτό. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν σήμερα συστήματα και προγράμματα επιδοτήσεων ε, που στηρίζονται σε κάποιες πολιτικές ε, κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τα προγράμματα αυτά στήριξης της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για τους συνεταιρισμούς θα πω ναι, αλλά ναι σε νέο τύπο συνεταιρισμών. Σας ζητώ συγγνώμη, λέει η αλλά θέλω να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Concord. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεταιρισμούς και συλλόγους ενώσεις γεωργών που να οδηγήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο λιανικό εμπόριο αλλά και στην ε, βελτίωση της παραγωγικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης γιατί εδώ η Επιτροπή παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην επιστική ασφάλεια. Ξέρετε όμως δεν αφήσατε στην δεύτερη ομιλήτρια αρκετό χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι λοιπόν πάρα πολύ σύντομη. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ε, επιστημιστικής ασφάλειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο και να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνοχή. Η διαδικασία για τους του 2020, τη στρατηγική 2020, που εμπεριέχει και τη συζήτηση για το θέμα αυτό, μας οδηγεί σε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι και στα πλαίσια των συζητήσεων που γίνονται στο G20 πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ εκείνων των θέσεων και των θέσεων που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ βλέπουμε ότι η θέση των μικροπαραγωγών δεν ε, είναι αρκετά εμφανής. Τώρα, για τα σχόλια που ακούστηκαν για τις τιμές, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι υψηλές τιμές δεν μεταφράζονται άμεσα σε περισσότερα κέρδη και έσοδα για τους γεωργούς. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ακούσαμε επίσης τις εταιρικέ σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι οι προτεραιότητες και οι στόχοι των παραγωγών οποροκυπευτικών είναι πάρα πολύ σημαντικές εδώ. Μιλήσατε επίσης για τις μονοκαλλιέργειες ή τις επιλογές για πολυμορφία. Το πιο βασικό είναι να υπάρχει βιώσιμη παραγωγή, οικολογική παραγωγή. Αύξηση της παραγωγής, ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι το 30% της παραγωγής καταστρέφεται, σπαταλάται. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν τόσο μεγάλη αύξηση της παραγωγής αν λάβουμε υπόψη μας και χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτό το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να πω. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour... Euh, Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε κυρία Σταμούλη και κυρία Ένεμα. Σας ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε που είναι πολύ χρήσιμες για τη δική μας τη δουλειά. Και ευχαριστώ και όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο που είναι και το τελευταίο για σήμερα. Ο συνάδελφός μας, Μάικλ Κάσμαν, έχει έρθει πλέον και θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του για την δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού. Μια διαδικασία έγκριση. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Το θέμα αυτής της αναθεώρησης το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και χαίρομαι που είναι εδώ ο Charles Rudy που διαπραγματεύτηκε την αναθεώρηση της συμφωνίας και με έχει ακούσει πολλές φορές να επαναλαμβάνω τα καλά μου λόγια για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει αλλά παράλληλα έχω αναφέρει πολλές φορές και τις ανησυχίες που έχουμε στο Κοινοβούλιο, ιδίως για το άρθρο 4. Δεν το αναφέρω ως κριτική, αλλά το αναφέρω ως στρατηγική για αυτά τα οποία προτείνω στο σχέδιο έκθεσης που βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να δείξουμε συνέπεια και συνοχή το Κοινοβούλιο είναι ε, συνεπές και θα πρέπει η Επιτροπή επίσης να είναι συνεπής όταν ζητάμε αναθεώρηση του άρθρου 8 και όταν μιλάμε για τη μη διακριτική μεταχείριση με βάση τον ε, γενετήσιο προσανατολισμό, διότι οτιδήποτε άλλο θα μας επανέφερε στους στίχους του βασιλιά Λίρ, όπου ο βασιλιάς Λίρ λέει στην κόρη του, που λέει ότι δεν τον αγαπάει, και της λέει τίποτα δεν θα βγει από το τίποτα. Θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη πολύ ψηλά. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο πάρα πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις παραμελούν και θυσιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδη δικαιώματα, το θέμα της πρόσβασης στα τρόφιμα, επισητιστική ασφάλεια, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, πολύ συχνά παραμερίζεται για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτές τις συμφωνίες που υποτίθεται ότι θα φέρουν οικονομικά ωφέλη για όλους, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν να το κάνουν. Λοιπόν, το άρθρο 95 τη συμφωνία Κοτονού είναι η νομική βάση. Το 2005 τον Ιούνιο έγινε η πρώτη αναθεώρηση και η δεύτερη αναθεώρηση το 2009 το Μάιο. Και ο κύριος λόγος ε, για την αναθεώρηση είναι το να διατηρήσουμε το χαρακτήρα της εταιρικής σχέσης μεταξύ χωρών ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι μια συμφωνία χωρίς προηγούμενο και θέλουμε να μπορέσει να προσαρμοστεί στις ε, διεθνείς σχέσεις των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για διάφορους τομείς μεγάλης σημασίας και για, τα δύο, και για τις δύο πλευρές. Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο και όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Οικονομική συνεργασία, εμπορικές ε, συμφωνίες, ε, τελικές σχέσεις, ανάπτυξη χρηματοδότησης, προγραμματισμός ε, της αναπτυξιακής βοήθειας και διαχείριση αυτής. θα πρέπει μέχρι τώρα να έχει επικυρωθεί από όλε τι χώρε ΑΚΕ και τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι έχει επικυρωθεί από όλε. Τώρα πάντω έχει φτάσει αυτή η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσει την συμφωνία του. Είναι το τελευταίο βήμα και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν λάθο να κάνουμε αυτό το τελικό βήμα χωρί να έχουν κάνει την επικύρωση αυτά τα κράτη-μέλη που ακόμη κολλησιεργούν. Ε, ο Επίτροπος Πίμπαλξ πιστεύει ότι εδώ έχουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Δίνουμε εμείς με την ε, επικύρωση ένα πολιτικό μήνυμα και προς τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τις χώρες ΑΚΕΑ. Υπάρχουν πολλά καλά σημεία στη συμφωνία. Ισχυρή διατύπωση όσον αφορά τους στόχους της ε, χιλιετίας, ε, επιστηστική ασφάλεια, συνέπεια στους στόχους μας, περιφερειακή ολοκλήρωση, ρόλος των ε, τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Έχω εκφράσει κάποιες ανησυχίες που τις έχουν εκφράσει και άλλοι, οι οποίες καλύπτονται στην έκθεση της κυρίας Ζολή του Δεκεμβρίου 2009. Όμως δεν ε, έχουν καλυφθεί όλα αυτά στο τελικό κείμενο, όπως είναι το θέμα της ε, επανεισδοχής των μεταναστών, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, γιατί αυτό είναι κέρια σημασία για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα φορολογικά στοιχεία. Και Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματα μέχρι τώρα έχει εκφράσει την επιθυμία του να τονίσουμε την αρχή ε, των μη διαπραγματεύσιμων ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το άρθρο 8 παράγραφο 4 για τον πολιτικό διάλογο δεν έχει αναδιατυπωθεί καταλήλω σύμφωνα με την επιθυμία του Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει μόνο τη διατύπωση του άρθρου 2 τη διακήρυξη των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι χώρε ΣΑΚΕ δεν ήθελαν να συμπεριληφθεί το θέμα του γενετήσιου προσανατολισμού και ίσω από μόνο το αυτό θέμα δεν θα ήταν ανησυχητικό. Αλλά σε 38 χώρε και η ομοφιλοφιλία παραμένει ε, ποινικό δίκημα. Κάτι το οποίο οδηγεί σε ε, κακή μεταχείριση των ατόμων που είναι ομοφιλόφιλοι ε, ε, τον οποίων ο γενετήσιος προσανατολισμός δεν είναι αποδεκτός. Ε, δεν θέλω να αναφέρω το Σέξπιρ για άλλη μια φορά, γιατί ε, δεν μπορούμε να δεχθούμε σιωπηλά αυτή την νομοθεσία που ποινικοποιεί τη σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ή του ότι κάποια άτομα επιλέγουν κάποια τέτοια κατεύθυνση. Έχω κάνει ε, συναντήσεις και με τον Αμπιπίλ από τα Ηνωμένα Έθνη και με τον Επίτροπο Πίμπαλξ και ε, πολλές φορές οι χώρες εκεί αρνούνταν να συζητήσουν ε, αυτό το θέμα του γενετήσιου προσανατολισμού και από τις χώρες και πρέσβεις μα είπαν ότι η τωρινή διατύπωση στο άρθρο 8 παράγραφο 4 δεν συμπεριλαμβάνει τον γενετήσιο προσανατολισμό. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα. Υπάρχουν οι καλές προθέσεις των διαπραγματευτών, οι καλές προθέσεις του Επιτρόπου και τα αιτήματα των εκπροσώπων των πολιτών που όμως δεν οδήγησαν πουθενά. Επαναλάβω τους στίχους από το Βασιλιά λέει ότι τίποτα δεν θα βγει από το τίποτα και γι' αυτό εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, αυτές τις ομάδες και να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα να μην θυσιάζουμε κάποια ανθρώπινα δικαιώματα και κάποια άλλα να τα σεβόμαστε γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο σε μια Ευρώπη των 27 μελών και των 500 εκατομμυρίων κατοίκων η Ευρώπη που γεννήθηκε από τη στάχτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όπου είδαμε ε, κρεματόρια σε ολόκληρη την Ευρώπη με βάση ε, κάποια διαφορά έγιναν όλα αυτά, διαφορά ατόμων έγιναν όλα αυτά τα εγκλήματα και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πιστεύω ότι πρέπει λοιπόν να, να θέσουμε τους όρους μας. Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για κάποια τμήματα της συμφωνίας που δεν αντικατοπτρίζουν τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούμε από όλα τα μέλη να αναθεωρήσουν τις μη ικανοποιητικέ ρήτρε σε μια τρίτη αναθεώρηση της συμφωνίας και εδώ συμπεριλαμβάνεται η σαφή σαμνία της μη διακριτικής μεταχειρίσης με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό στο άρθρο παράγραφος 8. Και όπως έλεγα προηγουμένως, στην έκθεση αυτή ασχολούμαι και με το άλλο θέμα που πιστεύω ότι πρέπει να ε, συζητήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και αν υπάρχουν ερωτήσεις... Σας υπόσχομαι ότι δεν θα παραθέσω όπως πάσματα από το Σέξπιρ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Εγώ μπορώ να σας πω καταρχήν ότι συμφωνώ με το άρθρο 8 παράγραφος 4 που προτείνεται με όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε και δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Δεν θέλει το λόγο η Επιτροπή. Θέλετε? Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω εν συντομία στον κύριο Κάσμαν. Εγώ δεν έχω να παραθέσω Σέξπιρ καταρχήν, αλλά Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στη συνεδρίασή σας, διότι όπως είπατε, είχα την τιμή να διαπραγματευθώ αυτή την αναθεώρηση συμφωνίας που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλα τα θετικά σημεία που υπογραμμίσατε διότι όντως επιφέραμε πολλά θετικά σε αυτή την αναθεώρηση που ξεκίνησε ως μια τεχνική προσαρμογή και κατέληξε να γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που τονίσατε τα σημεία στα οποία επιτύχαμε σημαντικές βελτιώσεις. αποτελούν μια ένδειξη όλα αυτά τα οποία διαπραγματευθήκαμε ότι αυτή η εταιρική σχέση είναι μια ζωντανή εταιρική σχέση που μπορεί να εξελίσσεται και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά και στο μέλλον. Δεν μπορέσαμε βέβαια να τα επιτύχουμε όλα και σημείωσα αυτά τα οποία μας είπε ο εισηγητής. Δεν ε, επιτύχαμε όλα όσα θα θέλαμε για την φορολογική διαφάνεια, για την κινητοποίηση των πόρων επιτόπου δεν επιτύχαμε όλα αυτά τα οποία θα θέλαμε. Βέβαια, ήμασταν και αρκετά απαιτητικοί έναντι των εταίρων μας από τις χώρες και Κάποια από αυτά τα οποία ζητούσαμε ίσως ήταν πολύ απαιτητικά. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν ότι αναθεωρήθηκε πλήρως το κεφάλαιο που αφορά το εμπόριο μπορεί να μην έγινε τεράστια πρόοδο, αλλά υπάρχει μια σημαντική διευκρίνηση, γιατί υπήρχε μια συμφωνία που δεν ήταν προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα, ενώ τώρα είναι και υπάρχουν σημαντικέ βελτιώσει εκεί. Τώρα, όσον αφορά κάποιε από τι επιφυλάξει του εισηγητού, γνωρίζουμε ότι δεν κατορθώσαμε να επιτύχουμε όλα αυτά που θα θέλαμε σε αυτά τα σημεία και παραμένουν στον κατάλογο των θεμάτων που θα πρέπει να επαναξεταστούν σε μια επόμενη αναθεώρηση. Τώρα, για το βασικό σημείο στο οποίο επιμείνατε, στο άρθρο 8, θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι ο πολιτικός διάλογος ε, δεν λειτουργεί. Τα θέτουμε τα ερωτήματα αυτά τα οποία σας απασχολούν στον πολιτικό διάλογο τα συζητήσαμε και μάλιστα βάλαμε τις κυβερνήσεις ε, να μπουν στη συζήτηση. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατα. Στην Ουγκάντα έγινε πολιτικός διάλογος με τον πρόεδρο για το θέμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο περνά παρατήρητο στις χώρες ΑΚΕ. Μπορεί να αρνούνται να συζητήσουν ε, αυτά τα θέματα όταν πρέπει να ακολουθήσουν μια κοινή θέση ενώ μεμονωμένα τα συζητάνε αυτά τα θέματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίσταση που είναι δύσκολο να ξεπεράσουμε όταν θέλουν ε, να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία. Σε μεμονωμένο επίπεδο όμως μας δίνουν διασφαλίσεις για την ομοθεσία που ενδέχεται να τροποποιήσουν και για το πώς αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα προβλήματα. Άρα στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Τώρα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ε, τα έχουμε συζητήσει. Γνωρίζετε ότι για την Επιτροπή είναι ξεκάθαρο ότι η τωρινή διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 4 επιτρέπει τη συζήτηση και μιλά συγκεκριμένα και για την διακριτική μεταχείριση για το γενετήσιο προσανατολισμό, γιατί έτσι εμείς ερμηνεύουμε το κείμενο των Ηνωμένων Εθνών. οι διαπραγματεύσεις σχεδόν να βάγισαν λόγω αυτού του σημείου, γιατί ήταν ένα σημείο ε, που δημιούργησε κλειδονισμού στις διαπραγματεύσεις και έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση τελικά αν θα σταματούσαμε τις διαπραγματεύσεις ή αν θα προχωρούσαμε. Και επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι το άρθρο 8 με την τωρινή του διατύπωση καλύπτει αυτό το θέμα και επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι είναι ένα θέμα που στο πολιτικό διάλογο συζητάτε, τελικά μονογράψαμε τη συμφωνία και την κλείσαμε, κλείσαμε τις διαπραγματεύσεις επ' αυτής της βάσεως. Αν συμφωνήσουν τα συμβαλόμενα μέρη για μια τρίτη αναθεώρηση, σίγουρα και αυτό το θέμα θα συμπεριληφθεί. Ακούσαμε το έτοιμά σα ε, και αναλαμβάνει αυτή τη, είμαι σίγουρος ότι θα αναλάβει αυτή τη δέσμευση η Επιτροπή. Προς το παρόν αυτό μπορώ να πω, γιατί ε, γνωρίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα και θα πρέπει να συζητηθεί. Και πέραν της τρίτης αναθεώρησης, αν το ξανασυζητήσουμε σε τρία ή πέντε ή έξι χρόνια για το τι θα γίνει μετά το 2020, αν έχουμε συμφωνήσει το 15, το 16, το 17, μέχρι να επικυρωθεί η συμφωνία θα έχει λήξει κιόλας. Σε πάση περιπτώσει θα πρέπει στο μέλλον να το συζητήσουμε και πολύ θετικό είναι ότι εσείς κινητοποιηθήκατε και μιλήσατε και με τους πρέσβεις των χωρών ΑΚΕ και μέχρι την επόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να υποφεληθούμε του χρόνου αυτού για να προετοιμάσουμε το έδαφος. Στις τελευταίες διαπραγματεύσεις οι χώρες ΑΚΕ μας είπαν ότι δεν έχουμε κοινή θέση επ' αυτού και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε γιατί δεν υπάρχει κοινή θέση και δεν θα συμφωνήσουν ποτέ οι χώρες εταίροι μα. Άρα ένα από τα βασικά διδάγματα που πρέπει να εξαχθεί από αυτό είναι ότι χρειάζεται δουλειά προετοιμασία, ούτω ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες συζητήσεις τη αναθεώρησης. Να μην υπάρχει δηλαδή απέναντί μας ένα μέτωπο, αλλά οι διαφορετικές θέσεις των χωρών και να μας επιτρέψουν να επιτύχουμε την πρόοδο που θα θέλαμε. Αυτά λοιπόν ως ε, προοπτική για το μέλλον. Ε, κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που μας ε, δίνει την σύσταση να δεχθούμε τη συμφωνία γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε και μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε περισσότερο αυτά τα θέματα, πράγμα το οποίο είναι επιθυμητό από όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύστασή σας να δοθεί η συμφωνία. Ελπίζουμε ότι θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Μάικελ γιατί αναφέρθηκε στη δική μου εργασία. Μίλησε για το τι πρέπει ακόμα να γίνει, τι πρόοδος είναι απαραίτητη και ότι δεν είμαστε ίσως ε, σε θέση να κυρώσουμε τη συμφωνία. ακούγοντα τον Μάικελ, συνειδητοποιώ ότι σήμερα ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 4, σας άκουσα και είπατε ότι το, συγγνώμη, το άρθρο 8.4. Το 8.4 καλύπτει και τις διακρίσεις κατά των ομοφιλοφίλων. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πρέπει να πούμε στην πλευρά ΑΚΕ και να το επαναλάβουμε. Όμως ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα είναι, επειδή εκείνοι έχουν αντίθετη άποψη, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο στο μέλλον να συμφωνήσουμε όσον αφορά αυτό το ε, αμφισβητούμενο σημείο. Δεν μπορούμε κάθε φορά να επανερχόμαστε με τις ίδιες θέσεις χωρίς να υπάρχει πρόοδος. Και θυμάμαι τη συνάντηση την οποία αναφέρθηκε και ο Μάικελ με τους ε, πρέσβεις των χωρών ΑΚΕ που μας είπε μας είπαν τότε ότι οι διακρίσεις κατά των ομοφιλοφίλων την έχουμε κληρονομήσει από τους, την εποχή της απεικιοκρατίας και ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε ταπεινοί όταν αναφερόμαστε στο θέμα αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, αυτή η σκόπελοι και ευχαριστώ τον Μάικελ, ο οποίος βεβαίως είναι πολύ ευαίσθητος για το θέμα αυτό και από τη μία δεν υποχωρεί ως προς την ουσία και συμφωνούμε σε αυτό, από την άλλη με ρεαλιστικό τρόπο ζητά από το Κοινοβούλιο την κύρωση της συμφωνίας. Θα πρέπει όμως να εκφραστούμε με σαφήνεια προς το άλλο ε, μέρος, προς την πλευρά και δηλαδή, ότι όπως είπε και ο Μάικλ θα πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των θέσεών μας. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορεί να ερμηνευθεί η μία και η άλλη θέση, γιατί υπάρχει περιθώριο ε, διαφορετικής ερμηνείας και θα πρέπει να το επεξεργαστούμε. Τέλος, ελπίζω μετά το 2020 θα υπάρξει μία ανανέωση της συμφωνίας ε, ίσως με άλλη μορφή, σίγουρα θα χρειαστούν ε, τροποποιήσεις, αλλά χρειάζονται πολιτικές δεσμεύσεις και ένα πολιτικό πλαίσιο έτσι ώστε να διασφαλιστεί το κεκτημένο και να μην εγκαταλείψουμε αυτό το πλαίσιο. Γιατί σαφώς αν κοιτάξει κανείς τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική, βλέπει ότι υπάρχει ένα κενό περιεχομένου πλαίσιο. Ευχαριστώ λοιπόν τον Μάικελ και θα τον στηρίξουμε στις συστάσεις του. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ποιος ζητάει το λόγο, κανείς. Ο κύριος Κάσμαν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη παρέμβασή σας και για την υποστήριξή σας. Ήσασταν απόλυτα συνεπείς στο θέμα αυτό, όπως και άλλα μέλη της Επιτροπής. Να πω στον Κλάους ότι η άποψή μου διαφέρει λίγο και θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό ως ομοφιλόφιλος άνδρας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι θα μπορούσε να έχω γεννηθεί εγώ στην Ουγκάντα ή στο Καμερούν ή την Ιγυρία ή κάποια από τις άλλες χώρες όπου αυτή τη στιγμή δεν έχει... Δεν σταματάει οι διακρίσεις, αυξάνονται. Είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο Μουσαβίνη, αλλά τι έγινε στο μεταξύ. Ο νόμος παραμένει. Η απειλή του νόμου αυτού στις ζωές των ανθρώπων παραμένει. Στην Ιγυρία δεν βελτιώνονται τα πράγματα, επιδεινώνονται. Στο Καμερούν το ίδιο. Ένα χρόνο αφού του σκοτώθηκε ε, ε, ο ε, ακτιβιστής στην Ουγγάντα. Έχει, έχει διωχθεί ο φόνος του. Όχι. Σας παρακαλώ, δείτε ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται που βασίζεται ακριβώς στον ακτιβιστή αυτόν στην Ουγγάντα. Μόνο στην Αφρική, όπου υπάρχει τόσος πόνος μπορεί να συνοδεύεται από τόσο γέλιο και αγάπη ε, το θέμα αυτό. Ε, ο Πάστορας λέει στην κηδεία του ότι ποτέ δεν ήξερα πώ ήταν ο Ντέιβιτ. Τώρα το ξέρω και θα καεί στην κόλαση ε, και οι φίλοι του, η οικογένειά του προσπαθούν να ανακτήσουν το φέρετρο το, του ανθρώπου που αγαπούσαν και ελπίζοντας ένας ε, αξιοπρεπής επίσκοπος να του ε, κάνει μια αξιοπρεπή ε, κηδεία, δείχνει ότι μια ζωή που θυσιάστηκε για το λόγο αυτό είναι μια ζωή παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Και... Γιατί λοιπόν είναι τόσο αναποτελεσματικό το άρθρο 8.4 για διάφορους λόγους. Πρώτον, λόγω της ε, αμοιβαίας ανησυχίας. Η ΑΚΕ λέει μπορεί να σας ανησυχεί αυτό εσάς ε, η διάκριση των ανθρώπων αυτών, αλλά εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου, άρα δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, άρα δεν υπάρχει καμία βάση πάνω στην οποία να μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Η ισχυρή εταιρική σχέση λέτε, εύχομαι να έχετε δίκιο, ε, λέτε ότι θα εξελιχθεί. Λίγα γνωρίζω αλλά λέω ότι αν δεν υπάρξει εξέλιξη διακυβεύεται η ύπαρξή μας ε, ως ε, άνθρωποι. Εγώ θέλω να βελτιώσω τη ζωή ανθρώπων σε ε, με διάφορα μέρη του κόσμου που συχνά ξεχνιούνται λόγω του χρώματος του δέρματός τους, της εθνοτικής τους καταγωγής ή επειδή είναι ομοφιλόφιλοι λεσβείες ή διαφυλετικοί. Και όλοι και τώρα που εκπνέει η συμφωνία, υπάρχει καλύτερος τρόπος ε, να αποσχοληθούμε από το να επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη για ανθρώπους που δεν ε, την έχουν. Γι' αυτό μπήκα στην πολιτική, στη δημόσια ζωή και γι' αυτό εκφράζω τις ε, ανησυχίες μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που ενδεχομένω να μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάσμαν. Και πριν κλείσουμε τη συνεδρία σα υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 21η Φεβρουαρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Μαρτίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτουμε τη συνεδρίαση και θα ξαναρχίσουμε αύριο το πρωί στις 10 και κλεισμένων των θυρών με μια ε, συζήτηση για το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας ε, και πιο πριν θα γίνει η συνάντηση των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ.